Είμαι ο ο μάλλον για τις ε, έκθεση για τις βασικές ε, τραπεζικές υπηρεσίες. Η Επιτροπή είχε ζητήσει μια τέτοια έκθεση σε ό,τι αφορά τη ε, πρόσβαση σε αυτού του ε, βασικού τραπεζικού οργανισμού, ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή είχε προτείνει σχετικό, σχετικό έκθεση. Η ΙΜΚΟ θα θέλαμε να διασφαλίσουμε ότι θα επηρεάσουμε την άποψη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Να ζητήσω λοιπόν από τον κύριο Κλούτε να, να κάνει μια εισαγωγή στο θέμα. Σα äh, Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να ξεκινήσω. Δεν είμαστε τόσο πολύ άριθμοι σήμερα το απόγευμα, αλλά δεν πειράζει. Νομίζω καταρχάς να κάνω κάποιες παρατηρήσεις για την έκθεση εν γέννη. Θεωρώ ότι η έκθεση, το είχα τονίσει και σε διάφορες περιστάσεις, αποτελεί μια καλή ευκαιρία για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για να παρουσιαστεί ως προσπιστής των δικαιωμάτων των πολιτών και των καταναλωτών. Νομίζω ότι τα τελευταία χρόνια ε, στα πλαίσια της κρίσης αυτό ίσως να μην προβληθεί αρκετά, γι' αυτό καλό είναι να το προβάλλουμε. Σε ό,τι αφορά τη σύσταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής υπάρχει και ένας φόβος που είχαμε και την προηγούμενο καλοκαίρι ότι το soft law, αυτό το ήπιο δίκαιο, δεν αποτελεί το κατάλληλο εργαλείο για να διασφαλιστούν τα δικαιώματα όλων των καταναλωτών στις τραπεζικές υπηρεσίες. Ε, νέα κράτη-μέλη είχαν ε, δηλώσει ότι δεν είχαν προγραμματίσει άλλες ε, δραστηριότητες, ακόμα και σε κράτη-μέλη που δεν είχαν εφαρμόσει την σχετική νομοθεσία. Η Βουλγαρία δήλωσε πολύ απλά ότι δεν πρόκειται να κάνει τίποτα παραπάνω. Άλλε χώρε οι οποίε δεν είχαν κάνει απολύτω τίποτα επίση δήλωσαν ε, μη πρόθυμε να προχωρήσουν σε άλλε δράσει και θεωρώ ότι αυτό είναι πραγματικά ντροπή. Θα πρέπει αυτά να διασφαλιστούν σε επίπεδο ε, κράτων μελών. Αναρωτιέμαι αν η επικουρικότητα είναι πραγματικά σωστό δρόμο. 231 τροπολογίες έχουν καταβληθεί για μια τέτοια μικρή έκθεση. Πολλέ από τις τροπολογίες είναι διευκρινιστική φύσεως. Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω συνάδελφοι. Κάποιες άλλες ε, προσθέτουν κάποιες επιπρόσθετες ενδιαφέρουσες ιδέες και κάποιες άλλες ε, δίνουν πιο πολλές πρωτοβουλίες στα κράτη-μέλη σε ό,τι αφορά την μεταφορά των πρωτοβουλίων. Εδώ νομίζω ότι θα υπάρχει μεγαλύτερη ανάγκη συζήτησης για το κατά πόσο θα πρέπει να υπάρχει προδιαγραφή από πλευράς Ευρωπαϊκής Ένωσης και σε ποιο βαθμό θα πρέπει να υπάρχει απόφαση από τα κράτη-μέλη. Για τις μεμονωμένες προτάσεις τώρα, για τα βασικά στοιχεία της πρότασή μου, σε ό,τι αφορά τους παρόχους και για το πεδίο εφαρμογής. Εγώ θα ήθελα το δυνατόν ευρύτερη βάση των παρόχων. Ανάλογα και με το αν πρόκειται για οργανώσεις, ενώσεις, credit unions, αλλά και άλλου είδους τράπεζες, όπως η τράπεζα των φαρμακοποιών, για παράδειγμα στη Γερμανία. Επί της αρχής ε, συμφωνούμε, αλλά άλλοι θέλουν να υπάρχουν ε, λιγότερες εξαιρέσεις, άλλοι θέλουν να δοθεί μεγαλύτερη περιθώριο ελιγμού στα κράτη-μέλη και είναι ότως ε, αληθές ότι τα κράτη-μέλη γνωρίζουν την κατάσταση σε κάθε μέλος καλύτερα, αλλά το τέλος, στο τέλος θα πρέπει να βρούμε μία λύση η οποία δεν θα είναι διακριτική προς τον καταναλωτή και δεν θα δημιουργεί ανισορροπίες σε ό,τι αφορά την παροχή τέτοιων υπηρεσιών. Αν διαπιστωθεί ότι σε κάποια κράτη-μέλη κάποιες τράπεζες ε, εκπροσωπούνται για παράδειγμα στην Ήπεθρο και υπάρχει ε, κάποια δυσαναλογία, θα πρέπει να υπάρχει ένας μηχανισμός εξισορρόπησης. Αλλά αυτό να το αποφασίζουν τα κράτη-μέλη με την ανάλογη εμπειρία. Το θέμα της πρόσβασης τώρα. Θα πρέπει να έχουμε δύο ομάδες ε, στόχο. Αυτή που δεν είναι τόσο ελκυστική για τις τράπεζες καταρχάς και δεν ε, μπορούν να ε, ανοίξουν τέτοιους λογαριασμούς, αλλά κατά δεύτερον θα πρέπει να ευκολυνθεί το διεθνικό άνοιγμα λογαριασμών. Αυτά θα πρέπει να ισχύουν κατά βάση για την Ευρωζώνη. Κάθε καταναλωτής που ανοίγει έναν ε, λογαριασμό σε κάποια χώρα θα πρέπει να έχει κάποια σχέση με αυτή τη χώρα. Αυτό το θεωρούμε σχετικά δεδομένο. Δεν θα πρέπει να δημιουργούμε εμπόδια για τις ομάδες στόχου που θα ανερούσαν την πρωτοβουλία, γιατί όλοι οι πολίτες έχουν ε, τέτοιο δικαίωμα επί της αρχής να ανοίξουν ένα λογαριασμό χωρίς να χρειάζεται αιτιολόγηση. Επίσης, σε κάποιες χώρες δεν μπορεί κανείς, για παράδειγμα, να συμβάσει εργασιακή σύμβαση, να νοικιάσει ένα διαμέρισμα, χωρίς να έχει τραπεζικό λογαριασμό και χωρίς να υποβάλει τα σχετικά τεκμήρια. Αυτό είναι ένα πρόβλημα. Αυτό δεν ισχύει σε όλες τις χώρες, αλλά σε κάποιες χώρες ισχύει. Αυτό να το λάβουμε υπόψη, λοιπόν. για την ψηφιακή ανάπτυξη σημαντική, αλλά δεν νομίζω ότι το να υπάρχει ε, ένας ε, λογαριασμός email, ηλεκτρονικός λογαριασμός, όπως προτείνεται στην τροπολογία 130, μπορεί να αποτελεί προαπαιτούμενο. Ε, επίσης, για την υποβολή τεκμηρίων στην τράπεζα, προτού ανοίξει ένα λογαριασμό. Τι γίνεται με τους πολίτες που δεν έχουν για παράδειγμα, ακριβούς λογαριασμούς. Δεν μπορεί να τους αρνούμαστε το δικαίωμα να ανοίγουν ένα κανονικό λογαριασμό πληρωμών. Προτείνονται πραγματιστικές και ρεαλιστικές προσεγγίσεις. Σε κάποια κράτη-μέλη δεν υπάρχει τέτοια υποχρέωση, αλλά αυτό μπορεί να αλλάξει στο εκείς μέλος μέλλον. Για το θέμα του κόστους. Αυτό είναι λίγο αμφιλεγόμενο. Έχει να κάνει με το γεγονός ότι στη Γαλλία δεν υπάρχουν και δεν ζητούνται τέλη για το άνοιγμα ενός ε, βασικού λογαριασμού. Γι' αυτό είχα προτείνει να μην υπάρχει χρέος για το άνοιγμα ενός λογαριασμού. Ωστόσο, το θέλω να είμαι δογματικός. Θεωρώ ότι είναι απαραίτητο να βρούμε μία σαφή θέση και τοποθέτηση. Κάποιοι άλλοι συνάδελφοι πρότεινα να υπάρχει κάποιο το στο στο τέλη. 10 ευρώ ενδεχομένως στο Βέλγιο. Το ποσό αυτό είναι 13 ευρώ ανά έτος. Ο κύριος ε, Λούτβι είχε πρότεινε 15 ευρώ. Θα πρέπει να συμφωνήσουμε αν επί της αρχής θέλουμε να επιτρέψουμε να υπάρχει τέτοια χρέωση και αν ναι, σε τι ύψος θα πρέπει να συμφωνήσουμε σε ένα κοινό ε, ποσό. Αυτό φυσικά δεν θα πρέπει να εμποδίσει άλλες χώρες να επιβάλλουν πιο χαμηλά τέλη. Αυτό είναι θέμα επικαιρότητα. Για τη λειτουργικότητα του λογαριασμού, εδώ δεν καταβλήθηκαν, δεν υποβλήθηκαν τροπολογίες, χαίρομαι γι' αυτό προβλέπονται κάποιες μικρές δυνατότητες. Ε, ωστόσο, υπερανάληψης η κυρία Γκέπχαρτ είχε προτείνει σε κάποιες ιδιαίτερες περιπτώσεις να υπάρχει μια πρόορη ε, ανάληψη και χρέωση του λογαριασμού. σε κάποιε περιπτώσει να υπάρχουν κάποιε καθυστερήσει που μπορεί να σχετίζονται με προβλήματα, με την τράπεζα του εργαζόμενου, για παράδειγμα, αν μεσολαβεί Σαββατοκύριακο, να υπάρχει περιθώριο ε, μια-δύο μέρε πίστοση για ενδεχόμενη υπερανάληψη. Εγώ θεωρώ ότι είναι κάτι το οποίο θα πρέπει να το εξετάσουμε, αλλά θα πρέπει να προσέξουμε. Αυτή είναι δική μου εμπειρία με τις τράπεζες ότι χρησιμοποιούν τέτοιες ευκαιρίες για να προχωρήσουν σε μακροπρόθεσμες πιστώσεις από τις οποίες κερδίζουν. Άρα είναι κάπως δύσκολη η ιστορία από... Ε, μάλλον, αλλά επί της αρχής θεωρώ ότι αξίζει τον κόπο να το κοιτάξουμε σε ό,τι αφορά την προστασία ε, για υπερχρέωση εδώ πέρα καταβλήθηκαν κάποιε τροπολογίε. Νομίζω ότι καλά θα κάνουν τα κρατημέλη να βρουν εδώ πέρα χρήσιμε λύσει για του πολίτε, γιατί θα πρέπει να υπάρχει μια Ευρωπα... Δεν είναι απαραίτητο μάλλον να υπάρχει μια ευρωπαϊκή βάση για τέτοιε πρωτοβουλίε. και νομίζω ότι και στο Βέλγιο υπάρχουν κάποιε ευλογέ λύσει και σε άλλε χώρε υπάρχουν εύλογε και λογικέ λύσει. Δεν πρέπει να υπερβάλλουμε. Αυτό για κάποιους είναι ένα πρόβλημα και θα πρέπει να δώσουμε το μήνυμα στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή ότι θα έπρεπε να δραστηριοποιηθεί στον τομέα αυτό προκειμένου τα κράτη-μέλη να καταλήξουν σε εύλογες λύσεις, σε υποχρέωση πληροφόρησης τώρα. Η πρωτοβουλία για τέτοιους βασικούς λογαριασμούς έχει νόημα μόνο αν ξέρουν οι πολίτες ότι υπάρχουν τέτοια μοντέλα. Η πρόταση Ludwig Schulung να προωθούνται αυτοί οι λογαριασμοί μέσω των υπαλλήλων των τραπεζών, θεωρώ ότι είναι ε, πολύ καλή και νομίζω ότι θα πρέπει να υπάρχουν και εγχειρίδια και να εξηγείται αυτός ο βασικός λογαριασμός ε, στα website και στα σχετικά ενημερωτικά φυλάδια από ό,τι καταλάβαμε από τις τράπεζες θα μπορούσε όλο το, όλο σύστημα να περάσει στο πλαίσιο της νομικής παροχής συμβουλών. Να το διευκρινίσουμε όμως ότι δεν πρόκειται για νομικά δεσμευτική παροχή συμβουλών εκ μέρους των τραπεζών. Αυτό είναι λίγο δύσκολο από πλευρά διατύπωση στα γερμανικά. Αυτό μας ε, επεσήμεναν οι εμπλεκόμενοι φορείς, αλλά νομίζω θα καταλήξουμε σε μια διατύπωση η οποία θα καλύπτει τι ανάγκες που πραγματικά ε, εννοούνται και να καταλάβει και ο τι δεν εννοείται, εν περιπτώσει. Τελευταίο σημείο για τις ε, εξοδικαστικούς συμβιβασμούς. Το συμπεριλάβουμε είναι μια πρακτική η οποία ήθιστε σε κάποιες χώρες. Υπήρξαν κάποιες τροπολογίες που εξέφραζαν ε, διστακτικότητες, κάποιες που ήταν υπέρ της ρύθμισης αυτής, κάποιες που ε, δήλωναν ότι δεν θα ήταν ε, σκόπιμο να συμμετέχει και η πλευρά του καταναλωτή. Θα πρέπει να κοιτάξουμε και το θέμα του κατά πόσο είναι ρυθμιστικό το θέμα αυτό για να δούμε πώς θα καταλήξουμε σε έναν ε, συμβασμό που να βγάζει νόημα. Εγώ θα πρότεινα να κοιτάξουμε ποιες είναι οι καλύτερες εμπειρίες που έχουμε από τα κράτη-μέλη και να βρούμε τι είναι το καλύτερο. Για τις προθεσμίες τώρα και ολοκληρώνω το σημείο αυτό. Σε ενισχυμένη συνεργασία βρισκόμαστε με την ε, Επιτροπή Προστασίας του Καταναλωτή. Για τις τροπολογίες θα πρέπει να λάβουμε υπόψη που προέκυψαν από την Επιτροπή ΕΜΚΟ και την Επιτροπή Προστασίας του καταναλωτή. 8 Μαΐου θα ψηφιστεί η γνωμοδότηση στην Επιτροπή αυτή και νομίζω ότι θα πρέπει να ολοκληρωθεί η συμβιβαστική διαδικασία, να υποβληθούν οι σχετικέ συμβιβαστικέ προτάσει, οι οποίε και να ψηφιστούν το συντομότερο δυνατόν μετά την 8η Μαου στην Επιτροπή Οίκων. Αυτά λοιπόν από πλευρά μου. Σα ευχαριστώ και πάλι, συνάδελφοι, για την ε, ε, καλή συμμετοχή και συμμετοχή και στις διαβουλεύσεις. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε κύριε Κλούτεν. Περνάμε τώρα στους κοιοδείς εισηγητές. Ο Γκέι Μίτσελ δεν είναι εδώ, θα περάσουμε στους σοσιαλιστές λοιπόν. Έχετε τον λόγο. Tack för ordet. Låt mig börja med att understryka att detta är en viktig fråga. Θα ήθελα να ξεκινήσω τονίζοντας ότι το ζήτημα αυτό είναι σημαντικό. Βλέπω να είναι πολύ μεγάλη αξία στο να έχουν όλοι οι καταναλωτές στην Ευρωπαϊκή Ένωση το δικαίωμα να ανοίξουν και να χρησιμοποιούν ένα βασικό τραπεζικό λογαριασμό. Αυτό θα είναι θετικό για πολλές ομάδες, θα παρέχει και καλύτερη λειτουργία στην ενιαία αγορά. Κοιτώντας τις τροπολογίες ε, καθίσταται σαφές ότι χρειάζεται να επιταχύνουμε τη διαδικασία, να την εστιάσουμε μάλλον τη διαδικασία, γιατί έχει διασπαρθεί με ένα σύστημα που λειτουργεί καλά ως βάση για τις τραπεζικές υπηρεσίε θα πρέπει να καταστεί καλέ, καθαρή αυτή η ανάγκη στις τροπολογίες. Δεν κάνουμε μια γενική έκκληση προς τα κράτη-μέλη για δράση. Πρέπει να δείξουμε ότι το παίρνουμε σοβαρά θα πρέπει να καταστήσουμε απολύτως σαφές τις υποχρεώσεις που θα πρέπει ή όχι να έχουν τα κράτη-μέλη. Πιστεύω ότι πρέπει να δώσουμε στα κράτη-μέλη περιθώριο λιγμών. Εγώ δεν είμαι ιδιαίτερα υπέρα, αλλά εάν πρόκειται να κάνουμε κάτι τέτοιο, θα πρέπει να καθορίσουμε σαφώς το πλαίσιο. Θα πρέπει να έχουμε συστήματα αλληλοσυνδεόμενα και διαδραστικά πολλά πλεονεκτήματα παρουσιάζει το να κάνουμε αυτό το σύστημα όσο το δυνατό πιο γενική φύσης και καθολικό. Όλοι οι φορείς θα έχουν την υποχρέωση να προσφέρουν ένα βασικό λογαριασμό και μια βασική σειρά προϊόντα θέλουμε να αποφύγουμε τον κίνδυνο του κοινωνικού στιγματισμού. Οι φορείς θα πρέπει να έχουν ως καθήκον και ως υποχρέωση να διαθέτουν, να καταστήσουν διαθέσιμα τέτοια είδη λογαριασμών. Θα πρέπει να προσέξουμε να μην προσφέρουμε κοινωνική υποστήριξη σε ορισμένες κατηγορίες ανθρώπων όσον αφορά το θα πρέπει να προσπαθήσουμε να μην αποκλίνουμε καμία κοινωνική ομάδα, να είμαστε δίκαιοι με όλους. Και το ποσό το οποίο θα βαρύνει τον κάθε καθαθέτη να είναι το ίδιο και χαμηλό. Κανένας δεν θα πρέπει να πληρώνει περισσότερο. Εξάλλου πιστεύω ότι θα πρέπει να εξειδικεύσουμε κάπως τα πράγματα για να ξέρουν όλοι αυτός ο βασικός τραπεζικός λογαριασμός, ποιο κόστος έχει. Και το τέλος είναι το ίδιο όλους. Θα πρέπει λοιπόν να γίνει σαφής αναφορά σε όλα αυτά τα θέματα. Τώρα, οι νομοθέτες ίσως έχουν πρόβλημα αν προτείνουμε κάποιο συγκεκριμένο ποσό. Και οι φορείς παροχής υπηρεσιών πολλές φορές ξέρουμε ότι καλύπτουν κάτω από την τελική τιμή την οποία δίνουν διάφορα επιμέρους ποσά. Δεν νομίζω ότι μπορούμε να μπούμε σε τόσο πολλές λεπτομέρειες. Η Επιτροπή θα πρέπει να ξέρει κατά μέσον όρο τι κοστίζει κάθε τέτοιος λογαριασμός, ώστε να μπορεί να παρέχεται, να αυτό ο λογαριασμό σε όλους. Θα μπορούσαμε να πούμε κατά μέσον όρο 55 ευρώ ετησίω. Και βεβαίω ο κάθε υποψήφιος καταθέτης θα πρέπει να πάει στην τράπεζα και να δει προσωπικά κάποιον που θα το εξηγήσει τι σημαίνουν όλα αυτά. Δεν μπορούμε να τα κάνουμε όλα μέσω ηλεκτρονικού υπολογιστή. Τώρα, αν κάποιο θέλει να πληρώνει λιγότερο, επίση θα πρέπει να πάει και να διαπραγματευτεί. Το βελγικό μοντέλο νομίζω ότι είναι το πιο κατάλληλο. Και θα πρέπει να προσπαθήσουμε όλοι να έχουν πρόσβαση σε έναν βασικό λογαριασμό. 15 ευρώ ενδεχομένως. ώστε να καλύπτονται οι βασικές ε, ε, υπηρεσίες που παρέχει η τράπεζα στον καταθέτη. Και αν βάλουμε κατά ανώτατο όριο ένα ποσό το οποίο δεν θα μπορεί να υπερβαίνει καμία τράπεζα, νομίζω ότι θα κάνουμε κάτι το θετικό. Διαφορετικά διευκρινίσουμε κάποια πράγματα, δεν θα μας βοηθήσει η νομοθεσία. Επίσης, αν πιστεύουμε ότι είναι ένα δικαίωμα για κάθε καταθέτη αυτός ο λογαριασμός θα πρέπει να δούμε πώς θα υπάρχει και η κάλυψη νομικής πλευράς. Κάποιες ιδέες που παρουσιάζονται στο έγγραφο της Επιτροπής και σε κάποιες τροπολογίες κατέθεσαν οι συνάδελφοι μου προκαλούν κάποια ερωτηματικά. Δηλαδή, πώς μπορεί να αποδείξει ένας καταθέτης ότι του αρνήθηκε η τράπεζα να του ανοίξει ένα λογαριασμό προσφέρονται κάποιες άλλες υπηρεσίες με λιγότερο κόστος. Εν πάση περιπτώσει, όσο περισσότεροι καταθέτες έχουν πρόσβαση σε τέτοιου είδους λογαριασμούς, τόσο μικρότερο θα είναι το κόστος. Θα πρέπει όμως να υπάρχει νομική κάλυψη για όλο τον κόσμο. Και υπάρχουν και καταθέτες που δεν μπορούν να ανοίξουν ένα τρέχοντα ε, λογαριασμό. Δεν έχουν δικαίωμα. Θα πρέπει όλες αυτές τις περιπτώσεις να τις καλύψουμε. Τώρα, αυτό το οποίο θα πρέπει να ισχύει και να διασφαλίζει τους καταναλωτές θα πρέπει να είναι ένας μηχανισμός γενικός που δεν θα οδηγήσει κάποιους ε, σε καταχρήσεις. Όλοι όμως οι καταναλωτές ε, πρέπει να έχουν το δικαίωμα να ανοίξουν ένα τρέχοντα βασικό λογαριασμό. άσχετο αν έχει κάποιος άλλες, ε, ε, άλλου τύπου καταθέσεις λογαριασμού. Τώρα μιλάμε εδώ για αυτό τον βασικό λογαριασμό. Νομίζω λοιπόν ότι θα πρέπει να υιοθετήσουμε την πιο απλή λύση και νομικά την πιο ασφαλή. Είδα ότι έχουν κατατεθεί πάρα πολλές τροπολογίες και είναι δύσκολο πολλές φορές να δούμε η κάθε μία από αυτές ποια ομάδα στοχεύει για να μην αποκλειστεί καμία κοινωνική ομάδα. Φοβούμαι ότι με κάποιες από αυτές αυτό συμβαίνει. Για να δώσω ένα παράδειγμα. Απαιτείται η ταυτότητα του δικαιούχου του λογαριασμού αλλά σε κάποιες περιπτώσεις θα πρέπει να υπάρχει και συνεργασία μεταξύ κοινωνικών υπηρεσιών και του φορέα που παρέχει αυτή την υπηρεσία, της τράπεζας, ώστε να καλύπτονται όλοι οι ενδιαφερόμενοι. Επίσης, θα πρέπει να δούμε τον τόπο κατοικίας του καταθέτη. Πολλές φορές Θα πρέπει λοιπόν να βρούμε και συμβιβαστικές λύσεις για να βοηθούμε. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ. Ο Φιλίπ Ντεμπάκερ είναι ο επόμενος. Ehm, ευχαριστώ, Πρόεδρε. Όπως και αναφέρθηκε και στην προηγούμενη συζήτηση, υποστηρίζει στι γενικέ γραμμέ και την γραμμή τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή και του εισηγητή σε ό,τι αφορά την πρόσβαση σε αυτέ τι βασικέ τραπεζικέ υπηρεσίε. Είμαι πεπισμένο ότι η κατοχή ενό τέτοιου τραπεζικού λογαριασμού είναι ε, σημασία για τη συμμετοχή στην κοινωνική ζωή σε ό,τι αφορά και την πτυχή τη κοινωνική συμπερίληψη, αλλά θεωρώ για να μπορεί κανείς να ε, αξιοποιήσει όλα τα πλεονεκτήματα της ενιαίας αγοράς. Γι' αυτό λοιπόν θεωρώ ότι κάθε κράτος μέλος θα πρέπει να υποχρεούται να παρέχει τέτοιες υπηρεσίες στην επικράτειά του. Ωστόσο, έχω κάποια σημεία στα οποία πρέπει να επιστήσω την προσοχή σας. Καταρχάς, σε ό,τι αφορά αν πρόκειται για νομοθετική ή μη πρωτοβουλία, δεν νομίζω ότι όλες οι χώρες ε, αντέδρασαν και ανταποκρίθηκαν στην πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Ο εισηγητής πριν από το τέλη του 2012 να υπάρξει νομοθετική πρωτοβουλία από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Σε περίπτωση ε, που δεν υπάρχει ανταπόκριση από το, Ευρωπαϊκό από το Συμβούλιο, θεωρώ ότι θα πρέπει να δώσουμε όντω ένα κίνητρο, αλλά θα πρέπει να ζητήσουμε πρώτα επιτακτικά στα κράτη-μέλη να λάβουν δράση μέχρι τα τέλη του έτου, να ζητήσουμε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή μέχρι τον Ιανουάριο του 2013 να καταρτήσει μία έκθεση για το πού ε, βρίσκονται τα πράγματα και αν δεν υπάρχει μέχρι τότε αυτή η εξασφάλιση των υπηρεσιών αυτών στην επικράτεια κάθε κράτου μέλου, να υπάρχει, να προτείνουμε στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή να, καταβάλει, να υποβάλει ε, νομοθετική πρωτοβουλία μέχρι τα Ιούλιο του 2013. Δεύτερο θέμα, ποιο μοντέλο θα πρέπει να χρησιμοποιηθεί για τέτοιες βασικές τραπεζικές υπηρεσίες. Εδώ θεωρώ ότι θα πρέπει να ακολουθήσουμε την αρχή της επικουρικότητας, γιατί υπάρχουν κάποιες χώρες που προβλέπουν ήδη τέτοιε δομέ και είμαι πεπισμένο ότι το τελικό αποτέλεσμα είναι αυτό που μετράει. Η πρόσβαση σε τραπεζικέ υπηρεσίε για κάθε πολίτη. Ο τρόπο με τον οποίο το διοργανώνουν αυτό τα κράτη-μέλη δεν θεωρώ ότι είναι τόσο σημαντικό και θεωρώ λοιπόν ότι στην έκθεση του Κοινοβουλίου δεν θα πρέπει να διαγράφονται υπερβολικέ ε, λεπτομέρειε για τα κράτη-μέλη. Γιατί σε χώρε όπου υπάρχουν τέτοιε ίδιε βασικέ ε, τραπεζικέ υπηρεσίε σε κάποιες τράπεζες ε, είναι η κεντρική τράπεζα αυτή που παρέχει τις υπηρεσίες αυτές ε, ή κάποια συγκεκριμένα ταμεία. Αλλά νομίζω ότι το σημαντικό είναι οι χώρες στις οποίες υπάρχει ήδη ένα τέτοιο σύστημα και το σύστημα αυτό έχει αποδεχτεί ότι αξίζει, δεν θα, πρέπει να τροποποιηθεί το σύστημα αυτό αναγκαστικά. Θα πρέπει να προσέξουμε επίσης και τους νέους παράγοντες στην αγορά τα prepaid solutions, οι κινητές, οι ε, θα πρέπει να ληφθούν υπόψη και σε μελλοντικές προτάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, γιατί αποτελούν καθημερινή πραγματικότητα. Ποιος θα πρέπει να μπορεί να χρησιμοποιεί τέτοιες βασικές τραπεζικές υπηρεσίες. Ε, αντίθετα με τον εισηγητή, πιστεύω ότι κάθε καταναλωτής ε, σε κάθε, θα πρέπει να μπορεί να ανοίξει λογαριασμό σε οποιαδήποτε βασικό λογαριασμό σε οποιαδήποτε χώρα. Μάλιστα, συγγνώμη, θα πρέπει να έχει κάποια σχέση με τη χώρα αυτή, είτε να είναι ε, φοιτητή, είτε να έχει κάποια άλλο σύνδεσμο, σύνδεση με το κράτος μέλος. Υπό την ευρία έννοια, αλλά να υπάρχει κάποια σχέση. Τι πρέπει να κοστίζει τώρα αυτή η βασική υπηρεσία ε, αρχικά προτείνει ο εισηγητής να μην υπάρχει κόστος. Ε, στη δική μου χώρα υπάρχει ένα κόστος 12 με 15 ευρώ. Και νομίζω ότι κάθε κράτος μέλος θα πρέπει να έχει το δικαίωμα να μην χρεώνεται οτιδήποτε για αυτές τις βασικές τραπεζικές υπηρεσίες, αλλά εν πάση περιπτώσει θεωρώ ότι θα πρέπει να σεβαστούμε τα διάφορα υφιστάμενα συστήματα. Και είμαι πεπισμένος ότι ποτέ δεν υπάρχει δωρεάν ε, προϊόν. Πάντα κάποιος πληρώνει τελικά το κόστος αυτό. Και νομίζω λοιπόν ότι θα πρέπει να προσέξουμε αν θέλουμε να τα διαμορφώσουμε όλα αυτά χωρίς ε, χρέωση. Το Ταμείο Αποζημίωσης. Αυτό συνδύεται με την προηγούμενη συζήτηση. Νομίζω ότι θα πρέπει να υπάρχει μια μικρή προμήθεια για ε, μια τέτοια υπηρεσία. Δεν είμαι υπέρ ευρωπαϊκής λύσης ε, και στο σημείο αυτό και ο εισηγητής αναφέρει ότι μπορεί αυτό να προκαλέσει ε, ανταγωνισμό μεταξύ των διαφόρων ιδρυμάτων, αλλά νομίζω ότι αν φροντίσουμε να γίνονται τέτοιε μικρέ πληρωμέ, δεν θα χρειάζονται καν τέτοιες αποζημιώσεις και δεν θα χρειαζόταν και σχετική γραφειοκρατία. Τελευταίο θέμα, το, η σημασία της ε, χρηματοπιστωτικής εκπαίδευσης, αν θέλετε, κατάρτισης, γιατί θεωρώ ότι πολλοί κόσμος που δεν έχει λογαριασμούς δεν ε, συνειδητοποιεί τι δικαιώματα έχει και τι μειονεκτήματα έχει και μια τέτοια λύση. Θα πρέπει λοιπόν ε, ο κόσμος αυτός να ενημερωθεί για τις δυνατότητες που έχει, αλλά θα πρέπει να προβλέψουμε και στην έκθεση και για τους ε, καταναλωτές εκείνους που δεν θέλουν να ανοίξουν ένα τέτοιο βασικό λογαριασμό. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ και αν υπομονώ και προσβλέπω στη μελλοντική συνεργασία με τον εισηγητή, ελπίζω να μπορέσουμε να καταλήξουμε σε ένα καλό συμβιβασμό, σε ένα τέτοιο σημαντικό θέμα για το οποίο συζητάμε επί εβδομάδες. Ευχαριστώ. Fine. Um, is on the... Μάλιστα, εκ μέρους του ECR, Ιβο Στρίτζακ. Ευχαριστώ κυρίε και κύριοι. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε που μου δίνετε το λόγο. Όσον αφορά αυτήν εδώ τη συζήτηση, έχω κάποια σχόλια. κάποια σχόλια, κάποιες ε, σημειώσεις που σχετίζονται με τις ε, τροπολογίες που έχω υποβάλει. Υπάρχει ένα συγκεκριμένο θέμα που εγώ τουλάχιστον προσωπικά δεν θεωρώ ότι είναι τόσο σημαντικό. Θα κάνω λοιπόν κάποιες γενικές φύσεις παρατηρήσεις αντίθετα από μερικούς άλλους συναδέλφους. Δεν πιστεύω ότι το ζήτημα του να έχει ή όχι ένα τραπεζικό λογαριασμό σημαίνει να αποκλείεσαι ή να μην αποκλείεσαι από την κοινωνική ζωή, από τη ζωή στην κοινωνία. Εγώ πιστεύω ότι κάτι τέτοιο δεν αληθεύει. Διότι προσωπικά και εσείς σίγουρα θα γνωρίζετε ανθρώπους στο περιβάλλον σας που κατά βάση δεν έχουν τραπεζικό λογαριασμό και δεν πιστεύουν ότι αυτό αποτελεί κοινωνική απαξίωση της ιδιότητάς τους ως πολιτών. Εάν προσπαθήσουμε να νομοθετήσουμε με κάθε κόστος ε, τέτοια νομοθεσία, πιστεύω ότι κάνουμε βήματα προς τη λάθος κατεύθυνση. Αν αμφίβολα, πιστεύω όλοι, κάθε ενήλικας που έχει κάποιο εισόδημα κάθε άτομο φυσικά θα πρέπει να έχει το δικαίωμα να ανοίξει ένα λογαριασμό σε οποιαδήποτε τράπεζα επιλέξει και όποια του κάνει ευχαρίστηση ε, ταυτόχρονα θα πρέπει να υπάρχει μια σωστά καθορισμένη σχέση μεταξύ μιας τράπεζας, ενός χρηματοοικονομικού ιδρύματος και ενός πελάτη αλλά αυτό θα πρέπει να λαμβάνει χώρα στο πλαίσιο μιας συμβατικής σχέσης ε, δηλαδή βάσει ενό συμβουλίου μεταξύ του χρηματοπιστωτικού οργανισμού και του καταναλωτή. Μόνο αυτοί, αυτές οι δύο οντότητε θα πρέπει, πιστεύω εγώ, βάσει του ότι είναι ε, αμοιβαία επωφελέ και για τους δύο, οι δύο μόνο αυτοί θα πρέπει να συμφωνήσουν για το πώς θα προχωρήσουν προς αυτή την κατεύθυνση. Έτσι λοιπόν, ε, εγώ το μελέτησα όλο αυτό και έριξα μια ματιά σε ορισμένες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης ε, βάσει του Ευρωβαρόμετρου στη Γερμανία το 2005 0,01 έως 0,06% των πολιτών δεν είχαν τραπεζικό λογαριασμό στη Ηνωμένο Βασίλειο το 2008 τα νοικοκυριά που δεν είχαν λογαριασμούς ήταν 3% και οι ενήλικες έρχονταν σε 2% στη Γαλλία και το Βέλγιο 10.000 άτομα που είναι ένας πολύ μικρός ε, αριθμός εάν το συγκρίνουμε με το συνολικό πληθυσμό στη Φιλανδία, Σουηδία και τη Δανία 100% των πολιτών διαθέτουν τραπεζικό λογαριασμό στη δική μου χώρα, στην Δημοκρατική της Τσαχίας. 89% των ενηλίκων έχουν τραπεζικό λογαριασμό. Στη Σλοβενία, για παράδειγμα, ωστόσο, μόνο το 15% δεν έχουν τραπεζικό λογαριασμό. Κοιτώντας λοιπόν αυτά τα μεγέθη, Πιστεύω ότι τα κράτη-μέλη το χειρίζονται μια χαρά ήδη από μόνα τους. Δεν χρειάζονται ευρωπαϊκή νομοθεσία για να αντιμετωπίσουν αυτό το ζήτημα. Βάσει όλων αυτών των στατιστικών στοιχείων και όλων αυτών των ποσοστών, εγώ προσωπικά δεν έχω την αίσθηση ότι, ότι υπάρχει κάποιο θεμελιώδες πρόβλημα πρόσβασης ε, στους βασικούς τραπεζικούς λογαριασμούς. Κατά συνέπεια, και αυτό είναι το ένα κομμάτι της τροπολογίας μου. Είναι μάλλον, σε αυτό αναφέρονται ορισμένε οι τροπολογίε μου. Θα ήθελα να συστήσω στην Κομισιόν να σεβαστεί την αρχή τη επικουρικότητα. Πραγματικά πιστεύω ότι τα κράτη-μέλη ξέρουν πώ να το χειριστούν. Πιστεύω ότι δεν πρέπει να του επιβάλλουμε ή να του πούμε τι πρέπει να κάνουν. Ε, η δεύτερη ομάδα των τροπολογιών μου βασίζεται στην πεποίθησή μου ότι θα πρέπει να υπάρχει μια σαφή σύνδεση μεταξύ μια τράπεζα χρηματοπιστωτικού οργανισμού και ενό πελάτη, ότι θα πρέπει να υπάρχει ένα συγκεκριμένο συμβόλαιο μεταξύ του. Αν θέλουμε να καθορίσουμε νομοθετικά πόσο θα πρέπει να σου κοστίζει να έχεις πρόσβαση σε τραπεζικές υπηρεσίες, κατά πόσο θα αφήσουμε του νομοθέτε να το καθορίζουν, ενώ φυσικά οι τιμέ διαφέρουν στις διάφορε χώρε συνάδελφοι αναφέρουν 12-15 ευρώ σε μια χώρα. Αυτό είναι ίσω το ελάχιστο ποσό σε ένα κρατός μέλο, Ωστόσο, το ίδιο ποσό μπορεί να είναι αρκετά υψηλό κόστο ε, σε μια άλλη χώρα. Κατά βάση όλες αυτές οι διαφορές τιμών είναι προφανείς ε, στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στις χώρες της και φοβάμαι ότι δεν έχουμε λάβει επαρκείς πληροφορίες ώστε να καθορίσουμε κάτι τέτοιο με ακρίβεια. Όλα αυτά σχετίζονται με τα κόστη. Πόσο πρέπει να πληρώνει κανείς για να ανοίξει ένα λογαριασμό ή τα κόστη που σχετίζονται με την εξυπηρέτηση των πελατών. Με τις υπηρεσίες προς τους πελάτες, ορισμένοι από εμάς για παράδειγμα, ο κύριος Σμιτ για παράδειγμα στην Νίμκο ε, σήμερα το πρωί ε, χρησιμοποίησε πολλά επιχειρήματα για να υποστηρίξει ότι θα πρέπει μέσα σ' άκρες να είναι δωρεάν εμείς ως νομοθέτες απλά δεν θα πρέπει να παρεμβούμε μεταξύ ε, στο μέσο αυτής της σχέσης μεταξύ των τραπεζικών ιδρυμάτων και των καταναλωτών αφετέρου. Πραγματικά δεν θέλω να εμπλακούμε σε αυτό τον καθορισμό των τιμών. Και ένα τρίτο θέμα. Το κατά πόσο αυτή οι βασικοί τραπεζικοί λογαριασμοί θα πρέπει να εντάσσονται σε ένα σύνολο υποχρεωτικών υπηρεσιών και αυτό θα βασιστεί επίσης, θα πρέπει να βασιστεί στις παραδόσεις των κρατών μελών. Ας μην προσπαθήσουμε να νομοθετήσουμε από ευρωπαϊκό επίπεδο λέγοντας ότι πρέπει να είναι υποχρεωτικό στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ή να λέμε ότι πρέπει απευθείας ότι ποιες υπηρεσίες πρέπει να περιλαμβάνονται, σε ποιους λογαριασμούς ε, και η τελευταία ομάδα των τροπολογιών μου αφορά κάτι άλλο. Δεν μιλάμε για νομοθεσία. Συχνά συζητάμε για κάτι το οποίο συνέβη στο παρελθόν, συνεπώς το γνωρίζουμε σήμερα. Ωστόσο δεν μπορούμε να προβλέψουμε τι θα συμβεί στο μέλλον και ποιες θα είναι οι εξελίξεις. Ε, έτσι λοιπόν θα πρέπει να είμαστε ε, αισιόδοξοι όσον αφορά την τεχνολογία γιατί είμαι σίγουρος ότι θα παρασχεθούν ε, υπηρεσίες οι οποίες θα καλύψουν αυτά τα κενά που παρουσιάζει η αγορά σήμερα θα υπάρξει κάποια μεταλλαγή αυτών των υπηρεσιών κατά κάποιο τρόπο. Αυτά είναι τα θέματα τα οποία περιλαμβάνονται και στις τροπολογίες μου που έχω υποβάλει. Ευχαριστώ πολύ για την προσοχή σας. Um, Πριν περάσω στον εισηγητή, θα αυτή τη συζήτηση και θέλω να κάνω ένα σχόλιο το 7% των πολιτών της Ευρωπαϊκής Κοινότητας που δεν χρησιμοποιούν τις τράπεζες ε, δεν αντιστοιχεί απαραίτητα σε ανθρώπους χαμηλού εισοδήματο. Αντιστοιχεί μερικές φορές σε ανθρώπους που φοβούνται ότι το να έχουν λογαριασμό σε μια τράπεζα είναι κάτι που δεν βρίσκουν κανονικό. Γι' αυτό πολλές χώρες ε, μετατρέπουν τα ταχυδρομεία τους σε κάποιο μορφή τραπεζών. Είναι αρκετά ενδιαφέρον ότι στην Αφρική, όπου το τραπεζικό δίκτυο είναι εξαιρετικά φτωχό και τα εισοδήματα είναι πολύ χαμηλά, έχουν βρει τρόπο να έχουν τραπεζικού λογαριασμού. Ο τραπεζικό λογαριασμό είναι απλά ο λογαριασμό του κινητού του τηλεφώνου και εταιρεία κινητής τηλεφωνίας τους επιτρέπει να κάνουν εμβάσματα, ε, αποταμίευση, γιατί είναι ευκολότερο για αυτούς να πάρουν ένα κινητό τηλέφωνο, να αποκτήσουν ένα κινητό τηλέφωνο το οποίο το θεωρούν απαραίτητο. Βρήκαν λοιπόν ένα τρόπο για τις βασικές τραπεζικές συναλλαγές τους σε ένα πολύ δύσκολο περιβάλλον όπως είναι η Αφρική. Αυτό λοιπόν θα μπορούσε να μας υποδείξει μια κατεύθυνση για να επιτύχουμε τους επιθυμητούς στόχους. Αυτό είναι απλά μια παρατηρήση μου, απλά και ας περάσουμε τώρα στον εισηγητή για να ολοκληρώσουμε τη ε, συζήτησή μας για αυτό το θέμα. Σας ευχαριστώ. Θα ήθελα να απαντήσω λίγο σε αυτά που είπε ο συνάδελφος Κυκλούνα. Πρόκειται και διαφορετικές κινήσεις ε, από την δεκαετία του 90 είχαμε την τάση να οικοδομηθεί ένα διαφορετικό οικοδόμημα γιατί υπήρχε διαφορά στο κόστος σε κάποιες τράπεζες. Κάποιοι, όλες οι τράπεζες έχουν αρχίσει να αποδυναμώνουν ε, τις υπηρεσίες αυτές. Γι' αυτό λοιπόν ε, θεωρώ ότι έχει νόημα η πρόβλεψη των χρόνων αυτών, αλλά εν πάση περιπτώσει πρόκειται για διαφορετικέ εξελίξει για αυτά που είπαν οι υπόλοιποι συνάδελφοι. Νομίζω ότι, κοιτάξτε, ε, έχετε δίκιο, συμφωνούμε νομίζω για τον Φίλιπ Ντεμπάκερ, νομίζω ότι μπορούμε να συμφωνήσουμε, θα βρούμε κάποια λύση για τη μορφή επικοινωνίας, ε, δεν αναφέρθηκα ιδιαίτερα στο θέμα αυτό, γιατί έχει να κάνει με το θέμα της ισότητας και της ανταγωνιστικής ε, ισορροπίας. Όσες τράπεζες έχουν εξαιρέσεις, θα πρέπει να έχουν ανταγωνιστικό πλεονέκτημα. Μας ενημέρωσαν ότι στο Βέλγιο ότι υπάρχουν κάποιες νομικές μορφές οι οποίες δεν εφαρμόζονται ωστόσο στην πράξη. Και η λύση με τα τέλη νομίζω ότι ρυθμίζεται στα πλαίσιο αυτό. Για αυτό που είπε ο Ιβο σε ό,τι αφορά τις τραπεζικούς λογαριασμούς ε, Λίγοι είναι αυτοί που δεν έχουν τραπεζικό λογαριασμό φυσικά. Αλλά διαβουλευτήκαμε και με τους καταναλωτές και κυρίως τους, στον κύκλο αυτό των ατόμων στην ε, Γερμανία υπάρχει μεγάλο πρόβλημα. Όταν ο κόσμος αυτός που δεν έχει τραπεζικό λογαριασμό και πριν από κάποια χρόνια μέχρι τη δεκαετία του 90, στο τέλος της δεκαετίας του 90 οι άνεργοι ε, βρίσκανε μια θέση εργασίας την οποία δεν μπορούσαν να πάρουν γιατί δεν είχαν τραπεζικό λογαριασμό. Τώρα πλέον έχει φυσικά αποσυμφορηθεί αυτή η κατάσταση, αλλά αυτό είναι το θέμα. Δεν μπορούμε να ε, υψώνουμε τέτοια εμπόδια για τον κόσμο. Ένα, για αυτό που άκουσα για τους ε, φοιτητέ, για τους μετανάστες, υπάρχουν κάποιοι οι οποίοι είναι πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και ζουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Θα πρέπει να προβλέψουμε και για αυτούς, αν θέλουμε μια Ευρωπαϊκή Ένωση για όλους τους πολίτες. Ακόμα και αν δεν είναι ο... Μάλλον το θέμα είναι η ενιαία αγορά, άρα δεν μπορώ να το αφήσω αυτό μόνο στο κράτη-μέλη. Πάντα τίθεται το θέμα ε, του ποιο πρέπει να είναι ο βαθμό τη επικουρικότητα, ποιο θα πρέπει να είναι ο βαθμό τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτό θα πρέπει να το έχουμε υπόψη μα. Αλλά νομίζω ότι ιδιαίτερα οι εμπειρίε σε ό,τι αφορά την ανακοίνωση του περσινού καλοκαιριού τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή μα καταδεικνύει ότι σε έναν τομέα που έχει να κάνει για, με πελάτες που δεν είναι πολύ ενδιαφέροντες για τις τράπεζες, εκεί δεν λειτουργεί η ρύθμιση στα κράτη-μέλη όπως θα έπρεπε να λειτουργεί. Γι' αυτό λοιπόν χρειαζόμαστε, θεωρώ, ευρωπαϊκή νομοθεσία να μην είναι υπερβολική, σύμφωνη, αλλά να θέτει ένα σαφές πλαίσιο για το τι αναμένουμε από τα κρατη Αλλά έχω την εντύπωση ότι σε κάθε περίπτωση θα βρούμε μια λύση. Σας ευχαριστώ και θα τα πούμε στις ε, επόμενες ημέρες ό,τι αφορά τις, στις, στα πλαίσια των συζητήσεων για την εξέβριση συμβασμών. Ευχαριστώ. Ε, ευχαριστώ κύριε Κνούντα. Ψηφοφορίες, όπως ήδη έχει λεφθεί, την Οίκον, 30-31 Μαΐου, τέλος Μαΐου δηλαδή, και πρόβλεψη ψηφοφορία στην Ολομέλη τον Ιούλιο. Φτάνουμε τώρα στο τελευταίο μας θέμα, που είναι αρκετά σύντομο. Τέλος, πάντων, λάθος έκανα, δεν είναι το τελευταίο θέμα. Πρόκειται για το δικό μου θέμα, που είναι γνωμοδότηση. Κύριοι λόγοι ανησυχία των επιχειρήσεων και των Ευρωπαίων πολιτών σχετικά με τη λειτουργία της ενιαίας αγοράς. Οι γνωμοδοτήσεις είναι κοινέ με άλλες επιτροπές. Στη δική μας δόθηκαν 20 από τους 26 κύριοι λόγοι ανησυχίες. Πρώτα απ' όλα, ε, τα θέματα, τα φορολογίες για διασυνοριακό εμπόριο. Το τρίτο είναι φορολογικά ε, θέματα, δυσκολίες στην χρηματοπιστωτική αγορά, πρόσβαση σε χρηματοοικονομικά και υποστηρικτικά μέτρα για την αγορά, και το τελευταίο αφορά το θέμα της απέτησης ΦΠΑ σε άλλες χώρες. Είπαν οι πολίτες λοιπόν της Ευρώπης ότι πιστεύουν ότι όλα αυτά είναι αρκετά επαχθή ως μέτρα. Εγώ εξέτασα τις διάφορες τροπολογίες που κατέθεσαν οι σκιώδεις εισηγητές και θα πρέπει να τονίσω ότι αυτή η γνωμοδότηση εστιάζεται όχι στις ανησυχίες όλων των Ευρωπαίων πολιτικών. Υπάρχουν πολύ περισσότερες από 20. Βρήκαμε τις 20, αν θέλετε, μεγαλύτερες αιτία ανησυχίας ε, και αφορά την ε, κινητικότητα των εργαζομένων, προβλήματα διασυνοριακά κτλ. Παρακαλώ λοιπόν τους και ηγητές να εμείνουν σε αυτά τα επιμέρους θέματα, διότι όντως δεν μπορούμε να εξετάσουμε προβλήματα που έχουν ε, οι πολίτες μας με συνήθι θέματα που αντιμετωπίζει ο καθένας στην Ευρωπαϊκή Ένωμα. Με κάποιες από τις τροπολογίες που έχουν κατατεθεί δεν έχω πρόβλημα. Θα μπορούσαμε να βρούμε ένα κείμενο αποδεκτό, συνενετικό, όπως φέρει πιν, το λέω αυτό για τον κύριο Ράπινγκ, για το κεφάλαιο και την φορολόγηση. Αλλά Υπάρχουν και άλλες τροπολογίες στις οποίες αναφέρεται η ενιαία εσωτερική αγορά σφαιρικά και λέγεται ποιες υπηρεσίες και οδηγία σχετικά με τις υπηρεσίες θα πρέπει να προχωρήσουν. Μάλλον καταδικάζουν τροπολογίες στην ενιαία εσωτερική αγορά διότι πιστεύουν ότι μεγαλύτερα προβλήματα δημιουργεί παρά επιλύει. Πιστεύω ότι τελικά υπάρχουν πολλές θετικές τροπολογίες τις οποίες θα μπορούσαμε να συζητήσουμε, αλλά πρώτα απ' όλα ας ακούσουμε τι έχουν να πούνε οι σκιώδεις εισηγητές. Η κυρία ε, Κονή, εκ μέρους του ΕΛΚ. Σοφία, έχει το λόγο. Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Πρόεδρε. Αγαπητοί συνάδελφοι, η έκθεση αυτή είναι ενδιαφέρουσα γιατί η ενιαία εσωτερική αγορά για πολλούς τομείς και για πολλά πράγματα είναι μια μεγάλη επιτυχία, αλλά βλέπουμε ότι ακόμη υπάρχουν προβλήματα και αδυναμίες και δυσλειτουργίες. Η οικοδόμηση ενιαίας εσωτερικής αγοράς δεν σημαίνει ότι θα πρέπει να υιοθετήσουμε εκατοντάδες οδηγίες κανονισμούς εναρμόνισης, αλλά να διαπιστώσουμε ότι στην καθημερινή ζωή των πολιτών τι ακριβώς λειτουργεί και τι ακόμη περισσότερο τι δεν λειτουργεί. Χαιρετίζω το γεγονός ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και ο Επίτροπος Μπαρνιέ ασχολούνται προσεκτικά με το θέμα της λειτουργίας ενίας εσωτερικής αγοράς. Η γνωμοδότηση του συναδέλφου Έντουαρτ Σικλούνα είναι ισοσκελισμένη. Δύο κυρία θέματα. Άρση των εμποδίων για την ε, ομαλή λειτουργία της ενιαίας εσωτερικής αγοράς και να υποστηρίξουμε την ανάλυση και την ε, ε, απασχόληση. Όπως λέει και ο Έντουαρτ και ο κύριος ε, Έπιν, θα πρέπει όντως τα φορολογικά εμπόδια να μπορέσουν να αρθούν. Όσον αφορά αυτά τα οποία είπε ο συνάδελφος Γκόκμαρ για την ανάπτυξη και την απασχόληση, συμφωνώ. Εγώ επέμεινα στην πρωτοβουλία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής δηλαδή υπέρ της κοινωνικής επιχειρηματικότητας και κυρίως για τον κανονισμό που θέλει να δημιουργηθεί ένα ευρωπαϊκό διαβατήριο για τα ε, επενδυτικά ε, κονδύλια τα οποία θα προωθούν σε τέτοιου είδους επιχειρήσεις. Ε, η έκθεση αυτή είναι έκθεση δική μου στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και βρίσκεται και μπροστά μας γιατί το επεξεργαζόμαστε εμείς και το Ευρωπαϊκό και το Συμβούλιο. Αυτό το διαβατήριο θα πρέπει να επιτρέψει να δημιουργηθεί ένα νέο επενδυτικό μέσον για τις επιχειρήσεις αυτές με τις οποίες ασχολούμαι εγώ, 10% του ποσοστού απασχόλησης και 11 εκατομμύρια πολίτες. Εδώ λοιπόν μπορούμε να έχουμε πολλές ελπίδες. Αυτό είναι το δικό μου το θέμα στην έκθεση αυτή, όπως σας είπα, διότι είχε σχέση με την έκθεση που κάνω εγώ και πρόκειται, επαναλαμβάνω, μια, για ένα πάρα πολύ καλό ε, κείμενο το οποίο κατέθεσε στα πλαίσια της γραμματότητας αυτής ο κ. Σικλούνα. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Δεν βλέπω να θέλει κανείς άλλο το λόγο. Άρα μπορούμε να συμπεράνουμε εδώ λέγοντας ότι η ψηφοφορία θα λάβει χώρα τέλος Μαΐου, 30 με 31 Μαΐου επίσης και η ψηφοφορία στην ε, επί της ουσίας αρμόδια επιτροπή 21 Ιουνίου και στην Ολομέλεια ψηφοφορία το Σεπτέμβριο.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 Είμαστε για 15 λεπτά πριν εξετάσουμε το επόμενο θέμα της ημερήσιας διάταξης.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 Uh, Συνεχίζουμε με το Ταμείο Κοινωνικής Επιχειρηματικότητας. Έχουμε 102 περίπου τροπολογίες για το θέμα αυτό. ECF, FMD. Δίνω το λόγο στην Σοφία Κονή να μας παρουσιάσει το θέμα της. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Αγαπητοί συνάδελφοι, πρόκειται για ένα θέμα το οποίο έχει προσελκύσει το πλήθος, αλλά πάση περιπτώσει, η ποιότητα, η σημασία και όχι ποσότητα. Θέλω να ευχαριστήσω σήμερα όχι τους παρόντες που είναι ελάχιστοι, αλλά όσους συναδέλφους κατέθεσαν τροπολογίες με στόχο να ενισχύσουμε, να βελτιώσουμε και να διευκρινίσουμε κάποια πράγματα στο κείμενο της έκθεσής μου. Συνεργαζόμαστε αυτή τη στιγμή όλοι για να μπορέσουμε να καταλήξουμε και στροπολογίες. Έχω πραγματικά εμπιστοσύνη τη συνεργασία και ελπίζω ότι οι συμβαστικές λύσεις θα μας οδηγήσουν σε μια πολύ καλή βάση συζητήσεις σε επίπεδο διαλόγου μεταξύ των τριών θεσμικών οργάνων. Όπως είπατε, 137 τροπολογίες που αφορούν κυρίως πέντε διαφορετικά θέματα. Πρώτα απ' όλα, ποιες είναι οι συνθήκες για να μπορέσει κανείς να πάρει την ετικέτα. Να κάνει επενδύσεις σε ποσοστό 70% στην κοινωνική ε, επιχειρηματικότητα. Κάποιοι όλο μειώσουν αυτό το ποσοστό σε 50% ή σε 30% με στόχο ευελιξίας και προσβασιμότητας. Άλλοι κατέθεσαν τροπολογίες όχι για τον αριθμό αλλά για την μέθοδο υπολογισμού διότι θέλουν να γίνουν αυτοί οι υπολογισμοί ώστε να καταλήγουμε σε μέσους όρους. Δηλαδή, έρχεται και Άστριντ, δηλαδή το 70% να μην απαιτείται συνέχεια στο ταμείο, αλλά κατά μέσον όρο να εξασφαλίζετε Η θέση μου είναι πολύ απλή. Το κατάφλι των 70% μου φαίνεται ότι είναι ισοσκελισμένο, διότι επιτρέπει να μην αποδυναμώνεται η ορατότητα, αν θέλετε, του τι κάνει αυτό το ταμείο στα πλαίσια της κοινωνικής επιχειρηματικότητας και κάτω από αυτό το κατόφλι θα είναι πάρα πολύ περιοριστικό. 70% λοιπόν νομίζω ότι είναι το κατάλληλο ποσοστό. Απ' την άλλη πιστεύω ότι θα πρέπει να διευκρινίσουμε την μέθοδο υπολογισμού, ένα μεσονόρο, της οποίας θα πρέπει να καθορίσουμε και τη διάρκεια που θα λάβουμε υπόψη για να κάνουμε αυτόν τον υπολογισμό. Εγώ φαντάζομαι ότι πέντε χρόνια είναι μια καλή περίοδος διάρκειας και ο στόχος αυτός, αν θέλετε, αιτιολογείται από την ε, νομική ασφάλεια που πρέπει να παρέχουμε. Τώρα, δεύτερος στόχος. Για τα ταμεία, τα επενδυτικά, 500.000 ευρώ. Για να μπορεί κανείς να έχει αυτή την ετικέτα, αν θέλετε. Όλα αυτά, βεβαίως, εάν γίνει σεβαστή η οδηγία IFM. Αυτή είναι η τροπολογία της Άστριντ. Και εγώ συμφωνώ μάλλον. Δηλαδή, ένα επενδυτικό ταμείο που είναι κάτω από 500, που δεν ξεπερνά τα 500 εκατομμύρια πριν να έχει την ετικέτα, εάν τα ξεπεράσει, παίρνοντας αυτή την ταυτοποίηση αν θέλετε, πρέπει να συνεχίσει να είναι επιλέξιμο. Σήμα. Σήμα. Λοιπόν, Τρίτο θέμα. Έτσι ε, θα πρέπει να διευρύνουμε, να είμαστε πιο περιοριστικοί όσον αφορά τον ορισμό της κοινωνικής επιχειρήσης. Ο στόχος είναι να μπορέσει να δημιουργήσει κοινωνικές επιπτώσεις θετικές. Μπορεί να ε, αποφέρει και σε κέρδη, αλλά αυτό θα πρέπει να είναι δευτερεύον, επικουρικό. Για να μπορέσει μια τέτοια επιχείρηση να είναι επιλέξιμη, θα πρέπει να παρέχει η αγαθά ή υπηρεσίες σε ευάλωτα ή περιθωριοποιημένα άτομα, μιλούμε εδώ για εργατικές κατοικίες, Φερρυπίν, ή για την ε, αλυσίδα αυτό κομμωτηρίων για ευάλωτα άτομα με πολύ φθηνές τιμές ή επιχειρήσεις και σας διαβάζω τον ορισμό μια επιχείρηση που χρησιμοποιεί μια μέθοδο παραγωγής υπηρεσιών ή αγαθών που είναι η υλοποίηση των κοινωνικών της στόχων. Πρόκειται για επιχείρηση λοιπόν η οποία απασχολεί άτομα με ειδικέ ανάγκες ή κοινωνικά ευάλωτα. Η πρότασή μου είναι ο ορισμός αυτός να διευρυνθεί κάπως. Για να καλύπτονται άτομα μη... που είναι αποκλεισμένα ή έχουν κάποιο μειονέκτημα και να αποδεικνύεται έτσι ότι κάνουμε μία πολιτική αλληλεγγύηση. Δεν θα ήθελα τώρα το σήμα αυτό να αποκλίνει από τον αρχικό του στόχο για αυτές τις επιχειρήσεις. Δεύτερο, τώρα, εάν θα πρέπει να διατηρήσουμε τον κατάλογο για τις ΜΜΕ ή όχι, να τον ξεπεράσουμε το κατόφλι κατά την άποψή μου αυτό θα πρέπει να το διαγράψουμε. Για να είμαστε πιο σαφείς και πιο ευέλικτοι. Οι εργατικές κατοικίες, Φερρυπίν, είναι επιχειρήσεις οι οποίες πολλές φορές ξεπερνούν την ε, ΜΜΕ. Κρίμα λοιπόν τέτοιου είδους ταμεία να μην ε, είναι ταμεία προσβάσιμα για αυτού του είδους τις εταιρείες. Γι' αυτό το διαγράψουμε και ενδεχομένως Ας μετρήσουμε το κατά κάποιον μπορούμε να έχουμε ένα άλλο κατόφλι όταν θα κάνουμε επανεξέταση σε τέσσερα χρόνια. Τρίτο σημείο. Επιλέξιμες τέτοιου είδους εταιρείε. Θα πρέπει να βρίσκονται στην Ευρώπη ή όχι. Αυτό το θέμα το συζητήσαμε αρκετά μεταξύ μας. Διότι μπορούμε να αποφασίσουμε. Να ευνοήσουμε μέσω αυτού του Ταμείου Κοινωνικής Επιχειρηματικότητας στην Ευρώπη επιχειρήσεις οι οποίες έχουν την έδρα τους στην Ευρωπαϊκή Ένωση και η ιδέα είναι το ταμείο αυτό να εξυπηρετεί μόνο τις επιχειρήσεις που βρίσκονται στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ώστε να δημιουργήσουμε έναν οικονομικό μοχλό για τις ευρωπαϊκές μας επιχειρήσεις και να βοηθήσουμε την κοινωνική επιχειρηματικότητα. Μπορούμε όμως να αποφασίσουμε να διευρύνουμε αυτό το ταμείο σε τρίτες χώρες. Σε επιχειρήσεις ε, κοινωνικής, σε επιχειρηματικότητας που εδρεύουν σε τρίτες χώρες. Θέλω όμως την άποψή σας. Τι πιστεύετε, πρέπει να ευνοήσουμε τις εταιρείες που βρίσκονται, τις επιχειρήσεις που βρίσκονται στην Ευρωπαϊκή Ένωση ή να δώσουμε αυτό το σήμα και σε επιχειρήσεις που βρίσκονται και σε τρίτες χώρες. Τέταρτη παρατήρηση. Άνοιγμα σε ιδιώτες επενδυτές. Πολλές τροπολογίες προτείνουν να μειώσουμε το κατόφλι των ταμείων σε 100 ή 50.000 ευρώ Και από 100 να πέσουμε πολλές φορές από 50 ή σε 30.000 ευρώ. Για να μπορέσουμε να το κάνουμε προσβάσιμο σε ιδιώτες. Μία άλλη λύση είναι η θέση μου. Να προβλέψουμε οι usage να επενδύουν σε τέτοιου είδους επιχειρήσεις σε ποσοστό 10% με το σήμα αυτό. Έχω την εντύπωση ότι αν προσφέρουμε αυτό το 10% στο Youth Seats, ευνοούμε τους ιδιώτες. Και ξέρουμε ότι υπάρχουν πολλοί ιδιώτες που θα ήθελαν να επενδύσουν 50.000 ευρώ για επιχειρήσεις κοινωνικής επιχειρηματικότητας. Σε τέτοιου είδους κεφάλαια κινδύνουν να επενδύσουν δηλαδή. Θα πρέπει λοιπόν να δώσουμε σε όλους αυτούς τους ιδιώτες την δυνατότητα να κάνουν μια τέτοια επένδυση σε ένδειξη αλληλεγγύης. Και τελικά, τελευταία παρατήρηση, ο θεματοφύλακας. Κατατέθηκαν τροπολογίες. Πρώτα απ' όλα προβλέπεται να υπάρχει ένα πολύ αυστηρό καθεστώς για τους Μια δεύτερη τροπολογία του συναδέλφου Όλε Σμιτ συνίσταται στο να έχουμε έναν τρίτο υπεύθυνο και μία, για τέτοιου μία, και μία τρίτη τροπολογία επιμένει στο ότι θα πρέπει να είναι υπεύθυνο ο διαχειριστής. Για μένα η συμβαστική λύση θα μπορούσε να είναι να υπάρχει ένας θεματοφύλας, κάποιος πιο light, ώστε να εξασφαλίσουμε μια κάποια ασφάλεια ορίζοντάς τον, αλλά έχοντας πάντα κατά νου την ευελιξία και κανόνες όχι πολύ επαχθείς. Πρέπει να σας πω ότι εγώ με μεγάλη υπερηφάνεια κατέθεσα, ε, ασχολήθηκα με αυτή την έκθεση που είναι πολύ ενδιαφέρουσα, το θέμα είναι πολύ ενδιαφέρον και το είπα και προηγουμένως όταν παρουσίασε την τροπολογία για την έκθεση Κλούνα. Πρόκειται λοιπόν για ένα τομέα, ο οποίο σήμερα, επαναλαμβάνω, περιέχει το 11% των ευρωπαϊκών επιχειρήσεων και 10 εκατομμύρια θέσεις απασχόλησης. Θα πρέπει λοιπόν εμείς στην Ευρωπαϊκή Ένωση να μεριμνήσουμε ώστε να εναρμονιστούν οι κανόνες, ώστε να μπορέσουμε πραγματικά να βοηθήσουμε αυτό το τομέα της οικονομίας. Ευχαριστώ. Thank you very much. Ευχαριστούμε πολύ. Με την άδειά σα, θα ζητήσουμε τον Ουλισμίτ επειδή έχει προηγούμενες δεσμεύσεις. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Το αεροπλάνο μου φεύγει σε μια ώρα. Ελπίζω ότι θα τα καταφέρω, ότι θα προλάβω, αλλά κανείς δεν ξέρει. Θα ήθελα να ευχαριστήσω την εισηγήτρια. Θεωρώ ότι η εκθεσή τη είναι εξαιρετική και ουσιώδου σημασία. Σημαντικό βήμα στο ευρύτερο φάσμα των επενδυτικών ταμείων στην ε, Ευρώπη. Έχω τέσσερις παρατηρήσεις. Θα προσπαθήσω να τις αναφέρω κατά προτεραιότητα. Η πρώτη αφορά τον θεματοφύλακα. Πιστεύω ότι θα πρέπει να εξετάσουμε το δεχόμενο ενός πιο ελαφρού καθεστώτος. Κατά την άποψή μου δεν θα πρέπει να συγκρίνεται με τα ταμεία εναλλακτικών επενδύσεων σε τέτοια περίπτωση αν κάνουμε τέτοια σύγκριση το όλο πλαίσιο γίνεται πιο περίπλοκο. Ελπίζω λοιπόν να καταφέρουμε να βρούμε μια συμβεβαστική λύση. Το δεύτερο που ήθελα να πω είναι ο ελάχιστος στόχος. Έχω μία τροπολογία για το 50%. Η πρόταση είναι 70%. Ελπίζω να μπορέσουμε να έχουμε έναν χαμηλότερο στόχο εδώ διότι και με αυτόν τον τρόπο τα ταμεία θα γίνουν ε, πιο περισσότερο αποδεκτά, τουλάχιστον κατά τη δική μου άποψη. Η τρίτη παρατήρηση που έχω να κάνω είναι ένα χρονικό όριο. Ελπίζω να μπορέσουμε να συμφωνήσουμε και σε αυτό. επειδή πιστεύω ότι να μην μπορούμε να υπερβούμε τα πέντε χρόνια είναι δύσκολο σε αυτού του είδους τα επενδυτικά ταμεία και ελπίζω και σε αυτή την περίπτωση να μπορέσουμε να καταλήξουμε σε μια εύλογη συμφωνία. Όλοι γνωρίζουμε ότι η Προεδρία της Δανίας ε, επιθυμεί να έχει κλείσει το φάκελο αυτό κατά την προεδρία της, κατά τη θητεία της. Τη τετάρτη παρατηρήσή μου αφορά τις καταχρήσεις και τις περιπτώσεις απάτης. Να μην χρησιμοποιούνται δηλαδή αυτά τα ταμεία για σκοπούς διαφορετικούς από αυτούς για τους οποίους προορίζονται. Αυτό αναφέρεται στο τροπολογισμούς 39 και 40 ότι πρέπει να αποφύγουμε οποιαδήποτε κατάχρηση σε περίπτωση που έχουμε ένα πιο ελαφρύ καθεστώς ε, δεν θα πρέπει να γίνεται κατάχρηση αυτού του καθεστώτος ε, και να ε, αξιοποιούνται χρήματα που κανονικά δεν αποτελούν κομμάτι αυτών των επενδύσεων. Κατά τα άλλα θεωρώ ότι η έκθεση αυτή είναι εξαιρετική. Όπως είπα είναι ένα βήμα προς σωστή κατεύθυνση διότι πιστεύω ότι λεφτά υπάρχουν και υπάρχουν και κονδύλια για να επιτύχουμε κάτι καινούριο στην Ευρώπη το ερώτημα που αφορά τις τρίτες χώρες ε, είναι λίγο πιο ευαίσθητο. Κατανοώ τα επιχειρηματά σας. Εγώ είμαι φιλελεύθερος, δεν μου αρέσουν πολύ οι φραγμοί. Διστάζω να πω λοιπόν ότι εδώ μιλάμε για μια ευρωπαϊκή αποκλειστικά κατάσταση. Αλλά αν εγώ ζητά ευελιξία εκ μέρου σας, ε, αξιότιμη κυρία, θα πρέπει και εγώ να επιδείξω ευελιξία στο πλαίσιο μιας αμοιβαιότητας. Θα ήθελα να ολοκληρώσω και ζητώ συγγνώμη και θα χρειαστεί να φύγω, ε, αλλά Όσα υπόθηκαν εδώ θα ε, συνταχθούν και εγγράφως από έναν από τους βοηθούς μας. Θα σας τα στείλω γραπτά ώστε να... Μάλλον θα λάβω γραπτά όσα θα πείτε εσείς εδώ συνεδρίαση. Και... Ευχαριστούμε. Περάμε στον κύριο Ελκαντράουι, εκ μέρους των Σοσιαλιστών. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Να ευχαριστήσω και τον εισηγητή την εισηγήτρια για την ε, εισαγωγή της και για το έργο της γενικότερα και λυζητώ συγγνώμη που έχασα ένα κομμάτι από την εισαγωγή τη. Αλλά αυτά που θα πω είναι μάλλον θετικά. Η κοινωνική οικονομία ασφαλώ και είναι ε, απαραίτητη και είναι ένα σημαντικό τομέα, το τονίσατε κι εσείς ε, και νομίζω ότι θα πρέπει να τραβήξουμε το ενδιαφέρον των επενδυτών. Αυτό είναι κάτι το απαραίτητο. Κάποιες παρατηρήσεις τώρα. Νομίζω ότι είναι σημαντικό να ορίσουμε σωστά το τι είναι η κοινωνική οικονομία. Θα πρέπει να είναι μια επιχείρηση καταρχάς που η οποία θα έχει ως ε, σκοπό προτεραιότητα να ε, πετύχει κοινωνικό αντίκτυπο και όχι τόσο πολύ την, ε, το κέρδος για τους μετόχους. Θα χρησιμοποιεί το κέρδος για την επίτευξη κοινωνικών στόχων. Και κάποιες ε, άλλες χαρακτηριστικά όπως διαφάνεια και τα λοιπά θα πρέπει να ε, υπάρχουν. Θα πρέπει να διευκρινιστεί όντως ένα τέτοιο ταμείο, τι ποσοστό επενδύει σε τέτοιες επιχειρήσεις κοινωνικής οικονομίας. Νομίζω ότι στο 70% για σε περίοδο 5 ετών είναι μια καλή βελτίωση σε σχέση με την αρχική πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και θα πρέπει να προσανατολιστούμε κυρίως ε, στον αντικτύπο στο ιστορικό της Ευρωπαϊκής Ένωσης και αυτό μου φαίνεται πάρα πολύ σημαντικό. Θα πρέπει να υποστηρίξουμε κυρίως τις επιχειρήσεις στο ιστορικό της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ποιος θα επενδύει σε ένα τέτοιο ταμείο. Αυτό θα πρέπει να το ορίσουμε σωστά. Εγώ υποστηρίζω να διευρύνουμε σε μια πιο μεγάλη ομάδα επενδυτών αν συνδεθούν όλα αυτά με μια κατάλληλη ε, προστασία των επενδυτών. Αυτά θεωρώ ότι πάνε μαζί και νομίζω ότι ο συμβιβασμό που προτείνει η εισηγήτρια προς αυτή την κατεύθυνση κινείται να το ελέγξουμε κατά πόσο να αποτελεί και από τεχνική άποψη την καλύτερη λύση, αλλά είμαστε θετικοί σε αυτά που προτείνεται για τον θεματοφύλακα. Εδώ είμαστε μάλλον ε, λιγότερο θετικοί. Θέλουμε ε, όσο το δυνατόν να υπάρχουν χαμηλότερα εμπόδια προκειμένου να χρησιμοποιήσουν όλο και πιο πολύ αυτή την ε, πρωτοβουλία. Θα πρέπει να το κοιτάξουμε λοιπόν αυτό, θα πρέπει να το σκεφτούμε λίγο καλύτερα. Αλλά εμείς θέλουμε ένα καθεστώς light, όσο πιο light γίνεται. Θα πρέπει να αναπτύξουμε όμως και εργαλεία και νομίζω ότι αυτό θα πρέπει να το πράξει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προκειμένου να προσμετράται ο κοινωνικός αντίκτυπος ε, των επενδύσεων. Και εδώ πέρα σας υποστηρίζω απόλυτα. Είναι νομίζω καλή προσθήκη αυτή και ασφαλώς για το ρόλο του Ευρωπαϊκού Εποπτικού Επόπτη. Συνοπτικά λοιπόν είμαστε πάρα πολύ θετικοί για την έκθεση και με τη γραμμή την οποία ε, προτείνεται θα υπάρχει ανάγκη να συζητήσουμε κάποια πράγματα αλλά νομίζω ότι θα λάβετε την υποστήριξη της ομάδας μου. Ευχαριστώ πολύ. Κυρία Λούλινγκ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ζητώ συγγνώμη την κυρία Κόνη γιατί έφτασα καθυστερημένη. Θα ήθελα να μου πείτε τι θα γίνει με τις δικές μου τις ε, τροπολογίες 53, 78 και 84. Γιατί εγώ είμαι τη άποψη ότι όντω θα πρέπει να είμαστε υπέρ του ανοίγματο προ τρίτε χώρες. Και στα πλαίσια της 53, της τροπολογίας μου δηλαδή, θα ήθελα να πω ότι θα ήθελα οι διαχειριστές έκτε και αυτοί που διαχειρίζονται τις ΟΣΕΚΑ να μπορούν και τέτοιου είδους ταμεία. Για την φορολόγηση τώρα των χρηματοπιστωτικών συναλλαγών δεν ψηφίσαμε τις τροπολογίες που είχαμε προτείνει κάποια από εμά. για να μην τις χάσουμε, τους χάσουμε αυτούς τους ΟΣΕΚΑ. Νομίζω ότι μπορούμε να κάνουμε κάποιες αλλαγές ακόμη στην Ολομέλεια. Διότι πιστεύω ότι οι συνάδελφοί που ήταν εδώ χθες δεν κατάλαβαν πάρα πολύ καλά ότι δεν θα πρέπει να επιβάλλουμε κυρώσεις στα ταμεία, τα οποία είναι ταμεία αποταμίευσης για κάποιους ιδιώτες καταθέσεις, καταθέτες μέσο και μακροπρόθεσμος. Διότι έτσι θα χάσουν εκατομμύρια ευρώ. Για να αρχίσουμε να φορολογούμε και να ξαναφορολογούμε και να ξαναφορολογούμε. Δεν ξέρω αν είπατε κάτι πριν όταν όσο δεν ήμουν εδώ. Απλώς εξηγήστε μου. Ευχαριστώ. Um, I understand the Commission would like to take the floor as well. Θέλει το λόγο. Ε, oui, merci, monsieur. Ναι, ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, ευχαριστώ κύριε Οκόνια και το σύνολο των μελών του Κοινοβουλίου που συνεδριάζουν εδώ σήμερα για αυτή τη συζήτηση και για τις τροπολογίες που παρουσιάστηκαν και που εκτιμάμε ε, κινούνται προς την κατεύθυνση βελτίωσης και εμπλουτισμού του κειμένου. Εν συντομία ήθελα να απαντήσω στο σημείο που παρουσίασε η κυρία Οκονιέ και που κατά την άποψή μου συνοψίζει σωστά το συζήτηση που θα κάνουμε επί της πρότασής σας πρώτα απ' όλα το ζήτημα των προϋποθέσεων λήψης του σήματος στο κατόφλιο του 70%, το γνωστό κατόφλιο. Συμφωνώ με το συμπέρασμα της κυρίας Σοκονιέ ότι το 70% μας φαίνεται ένα σημείο εξισορρόπησης μεταξύ της ανάγκης αφενός να διασφαλίσουμε ότι το σήμα κοινωνικής επιχειρηματικότητας δεν θα διαχυθεί, δεν θα διαμεριστεί παντού και ότι θα είναι ε, καθαρά, θα διακρίνεται καθαρά σε σχέση με άλλες προσφορές επενδυτικές παρέχοντας ταυτόχρονα την απαραίτητη ευελιξία για τη δημιουργία χαρτοφυλακίων ενδιαφέρων και ελκυστικών για τους επενδυτές. Επίσης αναφέρατε το ζήτημα του ενδεχόμενου χρονικού περιορισμού Αναφέρατε πέντε χρόνια πέραν του διαστήματος αυτού το Ταμείο θα πρέπει να έχει επενδύσει στο 70% που αναφέραμε. Η Κομισιόν δεν πρότεινε τέτοιο όριο. Θεωρούμε ότι έχει κάποια μειονεκτήματα όπως το ότι επιβάλλει στο τέλος, στο Ταμείο να επενδύει σε κοινωνικές επιχείρησεις που ίσως να μην είναι τόσο ενδιαφέρουσες και έτσι λοιπόν να αποτελεί καταλήτη επενδύσεων που δεν επιθυμούμε να ε, εγκαθιδρυθεί. Θα πρέπει να συνεχίσουμε τις συζητήσεις για αυτό το σημείο όσον αφορά τη σύνδεση με την οδικία AIFM είναι σημαντικό και σε αυτό το κοινοβούλιο και μεταξύ ορισμένων μελών υπάρχει βούληση για τα ταμεία που περνούν το κατόφλιο των 500 εκατομμυρίων να συνεχίσουν να χρησιμοποιούν το σήμα. Είναι απολύτως εύλογο αυτό. Αυτό θα έχει ίσως ε, ως συνέπεια το να πρέπει να ρυθμίσουμε κάποια τεχνικά ζητήματα, κυρίως όσον αφορά την αλληλεπίδραση μεταξύ των υποχρεώσεων της οδηγίας AFM που ε, προστίθενται στι υποχρεώσει του κανονισμού που συζητάμε σήμερα. Πιστεύω ότι αυτό το σημείο θα μπορούσαμε να το συζητήσουμε περαιτέρω και σε περισσότερο βάθο. Το ζήτημα του ορισμού κοινωνικός είναι σημαντικό. Η Κομισιόν προσπαθεί να κοινοτομήσει σε αυτό το τομέα, προτείνοντα έναν ορισμό, ο οποίο σχετίζεται με τον ορισμό που είχαμε προτείνει στην ανακοίνωση για την κοινωνική επιχειρηματικότητα. Εδώ υπάρχει περιθώριο προσαρμογής του κειμένου, έχουμε σημειώσει και τις πιθανές δυσμένες επιπτώσεις που θα μπορούσε να έχει αυτός ο ορισμός σε ορισμένες προσφορές επενδύσεων όπως την κοινωνική στέγη που αναφέρατε για παράδειγμα. Ένα άλλο σημαντικό και ευαίσθητο σημείο είναι η θέση στην Ευρώπη, η στην Ευρώπη των επιλέξιμων επιχειρήσεων. Δεν θέλουμε εμείς να θέσουμε τέτοιο περιορισμό για δύο λόγους. Πρώτον, στο χρηματοοικονομικό ρυθμιστικό μας πλαίσιο δεν έχουμε τέτοιο τύπου περιορισμό όσον αφορά τις ε, δυνατότητες επένδυσης. Μιλάμε για ελεύθερη διακίνηση κεφαλαίων αλλά και για λόγους που σχετίζονται με το γεγονός ότι ορισμένοι ιδρυτές κοινωνικών ταμείων θα ήθελαν να έχουν τη δυνατότητα σε επενδύσεων όσο πιο, το δυνατόν πιο ευρύες ώστε να μπορούν να συνθέτουν χαρτοφυλάκια ελκυστικά και εντός ε, χρονοδιαγραμμάτων συμβατών με το γεγονός ότι έχουμε να κάνουμε μια σχετικά νέα αγορά στην Ευρώπη και με μια προσφορά επενδύσεων σε κοινωνικές επιχειρήσεις που ίσως να μην είναι τόσο ε, άφθονη όσο θα πίστευε κανείς εκ των προτέρων. Αλλά δύο σημεία, το επίσης σημαντικό ερώτημα της πρόσβασης των ταμείων στους ε, ιδιώτες επενδυτές ε, ούτε εμείς, εμείς δεν θέλαμε να προτείνουμε κάτι τέτοιο παρότι εκτιμούμε ότι σε μεσοπρόθεσμα ο στόχος είναι εύλογος ωστόσο θεωρούμε ότι δεν είμαστε έτοιμοι για να προτείνουμε ένα κανονιστικό πλαίσιο σε αυτόν τον τομέα που ταυτόχρονα θα επιτρέπει να υπάρχει μια ε, προσφορά ελκυστική που θα υπόκειται σε ένα ελαφρύ κανονιστικό πλαίσιο αλλά και που παράλληλα θα μπορεί καθώς θα έχουμε να κάνουμε με ιδιώτες επενδυτές να εξασφαλίζει απαραίτητη προστασία. Σημειώσαμε την πρόταση της κυρίας Σοκόνια να ανοίξουμε ε, τις επενδύσεις των ταμείων στα ε, USATS. γιατί επαναλαμβάνω ότι ο στόχος είναι εύλογος, αλλά οι συνέπειες όσον αφορά την προστασία των επενδυτών, όσον αφορά την ενημέρωση των επενδυτών, κατά την απόψή μας ε, δεν είναι επαρκώς ενδιαφέρουσες για να προχωρήσουμε προς αυτή την κατεύθυνση. Ένα τελευταίο σημαντικό σημείο, το σημείο του θεματοφύλακα, είναι ένα σημείο το οποίο συζητήθηκε σε μεγάλο βαθμό στο Συμβούλιο η Κομισιόν θεώρησε ότι δεν ήταν σκοπό στην πρότασή της να περιλαμβάνεται μια υποχρέωση καθορισμού θεματοφύλακα. Έχουμε δείξει μια ανάλυση κόστους ωφελών και εκτιμήσαμε ότι το κόστος στο οποίο θα συνεπάγεται η υποχρέωση ε, θεματοφύλακα υπερβαίνει υπερβολικά τους κινδύνους ε, στοιχείων του ενεργητικού ή μη ε, των κανονών που θα μπορούσε να περιορίσει εν λόγω θεματοφύλακας. Θα αναφέρω δύο σημεία. Το πρώτο είναι ότι ίδια, ο ίδιος ο τομέας και αναφέρομαι τώρα στην ακρόαση που έλαβε χώρα στο πλαίσιο αυτής τη της Επιτροπής η οποία δεν ήταν ιδιαίτερα υπέρ του ορισμού θεματοφυλάκων και το δεύτερο είναι επίση σημαντικό να γνωρίζουμε γιατί μιλάμε όταν μιλάμε για θεματοφύλακα. Είναι σημαντικό η συζήτηση που κάνουμε επί αυτού του θέματος ε, να αναγνωρίζει καλά τόσο τους κινδύνους όσο και τα ε, καθήκοντα που θα θέλουμε να έχει ο θεματοφύλακας. Πρόκειται για κινδύνους απώλειας στοιχείων ενεργητικού, κινδύνους μη τήρησης των κανόνων που εφαρμόζονται στο Ταμείο, για τους οποίους θα μπορούσε να αποδειχθεί χρήσιμο σε ένα εξωτερικό θεματοφύλακας. Ε, αυτά τα στοιχεία θα πρέπει να τα έχουμε στο νου όταν συζητάμε για αυτό το θέμα. Θα σταματήσω εδώ κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστώ που μου δώσετε το λόγο. Σα Um, will... ευχαριστώ. Να στραφούμε προ την κυρία Οκόνη, την εισηγήτρια, για να συνοψίσει. Merci, Monsieur le Président. Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε, αγαπητοί συνάδελφοι. Άκουσα όλες τις αναλύσεις που έκαναν οι συνάδελφοι. Θα ήθελα πάρα πολύ σύντομα να τους πω ότι όντως θα συνεχίσουμε να συνεργαζόμαστε με επικοδομητικό πνεύμα έτσι όπως το κάνουμε και διάρκεια όλων των συζητήσεων. Ο κύριος Αλκαντράουι μίλησε για τον ορισμό της κοινωνικής επιχείρησης. Ξέρω ότι αυτό όντως το θέλετε και λάβαμε υπόψη τη δική σας πρόταση και όντως πιστεύω ότι θα οδηγηθούν προς αυτή την κατεύθυνση. Ο κύριος Όλε Σμιτ θέλει να έχουμε ένα λιγότερο επαχθές, πιο ελαφρύ καθεστώς. Δεν θελήσαμε να συγκρίνουμε ή μάλλον δεν ε, θελήσαμε να βασιστούμε στον κανονισμό που υπήρχε για τους ΟΣΕΚΑ. Ε, θα πρέπει όμως όλοι μαζί να τα κοιτάξουμε αυτά τα θέματα σε συνεργασία. Όσον αφορά την τροπολογία του αναφέρεται στο κατόφλι του 70% που θα ήθελε να κατέβει στο 50% ο Λεσμίτ. πρόκειται για σημεία τα οποία θα τα συζητήσουμε μαζί. Άστριντ, ήδη λάβαμε υπόψη κάποιες από τις τροπολογίες σας και είχα προβλέψει ούτως ή άλλως να έρθω σε επαφή μαζί σας, ώστε διμερώς να μπορέσουμε να συζητήσουμε και να διαπραγματευτούμε κάποιες από τις πολύ ενδιαφέρουσες προτάσεις σας. Αγαπητοί Άστριντ, Σα συγχωρώ τα πάντα. Ακόμη και την καθυστέρηση, γιατί ξέρω ότι είσαστε πάρα πολύ απασχολημένοι. Δεν υπάρχει πρόβλημα. Αυτό που θα ήθελα να πω είναι ότι όντω εγώ εκτίμησα όλους ιδιαίτερω το κλίμα μέσα στο οποίο διεξήχθηκαν το σύνολο των διαπραγματεύσεων. Θα συνεχίσουμε να συνεργαζόμαστε. Θα Ήθελα να ευχαριστήσω την Ευρωπαϊκή Επιτροπή όλους ιδιαίτερω για την πρόταση κανονισμού, την ποιοτική αυτή πρόταση που υπέβαλε. Να ευχαριστήσω την ε, και Προεδρία και το Συμβούλιο, καθώς και τη γραμματεία της ΕΚΟΝ, με την οποία με πολύ μεγάλη ευχαρίστηση εργάζομαι και το σύνολο των συναδέλφων για το καλό κλίμα το οποίο μπορέσαμε να δημιουργήσουμε στη συζήτηση αυτής της έκθεσης. Ευχαριστώ. Regarding Προθεσμία κατάθεση τροπολογιών τέλος Μαΐου και πάλι 30-31 και ολομέλεια ή του Ιουλίου ή του Σεπτεμβρίου. Αλλά αργότερα θα έχετε πιο πολλές διευκρινήσεις. Τώρα, μία πολύ παρεμφερής έκθεση με αυτή που έπρεπε να συζητηθεί συγχρόνως. Αλλά αποφασίσαμε να τις κάνουμε διαδοχικά. Ταμείο κινδύνων ε, κεφαλαίων κινδύνου. Πάλι έκθεση του κυρίου Λάμπερτς με πολλές τροπολογίες. Ο ίδιος ο Φιλίπ να το θέμα. Ευχαριστώ πρόεδρε. Α, θα μιλήσω γαλλικά αφού είναι εδώ και η Σοφή. Διότι νομίζω ότι οι πολυπληθοί συνάδελφοι στην αίθουσα καταλαβαίνουν τα γαλλικά. Ευχαριστώ, συγγνώμη που άργησα, αλλά πηδάω από τη μια συνεδρία στην άλλη. Δεν πρόκειται για δύσκολο φάκελο σε σχέση με άλλα. Δεν νομίζω ότι μας δημιούργησε μεγάλο φόρτο εργασίας, ούτως ή άλλως ήταν πάρα πολύ επικοδομητική συνεργασία. Συνεργασία στο Στρασβούργο συζητήσαμε οι μεταξύ μας. Ένα σημείο που είναι ε, κρεμές ακόμη, θα αναφέρω τώρα, στα πλαίσια τις δημιουργίε αυτού του ταμείου θα πρέπει όπως κάναμε και για το IFM και όπως κάνουν μια-δυο χώρες Ευρωπαϊκής Ένωσης να έχουμε πάντα έναν ε, θεματοφύλακα. Αν έπρεπε να ψηφίσουμε Για λόγους απλοποίησης, τι θα λέγαμε, ότι έχουμε να κάνουμε εδώ με ένα καθεστώς εξαίρεση σε σχέση με τα IFM. Θα πρέπει λοιπόν να είμαστε πάρα πολύ απλοί σε αυτό που κάνουμε. Καταλαβαίνω το επιχείρημα κάνουμε. Όλα εξαρ... θα εξαρτηθούν βεβαίως από τα διάφορα επιχειρήματα τα οποία ε, θα μου παρουσιάσουν η Γαλλία και το Λουξεμβούργο που είναι υπέρ. Θα δω ανάλογα με τι θα πούν λοιπόν. Επίσης θα μπορούσαμε να πούμε ότι θέλουμε να προστατεύεται ο καταναλωτής. Ναι, εδώ όμω μιλούμε για ένα ελάχιστο ποσό 50.000 ευρώ. Μιλούμε λοιπόν για καταναλωτές που έχουν μια κάποια οικονομική επιφάνεια και μπορούν να κρίνουν κατά κάποιο τρόπο αν υπάρχει κίνδυνος συμμετοχής σε τέτοιου είδους εταιρείες τις οποίες θέλουν να επενδύσουν. Εγώ πιστεύω ότι πρέπει να μείνει ανοιχτό το θέμα και αν δεν το συμπεριλάβουμε στο κείμενο με τα άρθρα, να πούμε σε μία ρήτρα αναθεώρησης αυτό είναι ότι αυτό είναι ένα θέμα στο οποίο θα πρέπει να ψήσει την προσοχή της η Επιτροπή κυρίως αν στο μέλλον θέλουμε να μειώσουμε το κατόφλι αυτό. Δηλαδή, εάν θέλουμε ένα καθεστώς όπου θέλουμε να προσελκύσουμε μικρούς επενδυτές, το κρατήσουμε. Ούτω ή άλλω, εγώ δεν έχω διαμορφώσει την ε, δική μου θέση. Θα δούμε ποια είναι η άποψη της πλειοψηφία και τις επόμενες ημέρες και διάρκεια της ε, τουρκουάζ εβδομάδας θα δω τι θα πάρω. Στα υπόλοιπα ε, θέματα είπαμε ότι όντω τα δύο πρώτα χρόνια θα πρέπει να υπάρχει ευελιξία πριν να μπορέσουν τα ταμεία αυτά να επενδύσουν τα κονδύλια τους κατά 70% σε ε, επιλέξιμες επιχειρήσεις. Οι επιχειρήσεις που κάνουν καινοτομία στο... θα πρέπει να συμπεριληφθούν όντως στον ε, τομέα αυτό, τον χρηματοπιστωτικό είδαμε καινοτομίε, αλλά όχι πάντα προς σωστή κατεύθυνση. Άρα είπαμε ότι για τα καινοτόμα σχέδια θα πρέπει να έχουμε εταιρείε ε, κεφαλαίων κινδύνου που να μην είναι σχεδόν αμυγός ε, χρηματοπιστωτικές. Επίσης, διαγράφει αναφορά στο closed end fence, ώστε να μην γίνει ακαμπτό το σύστημα ή δισκαμπτό και ο ορισμός των ε, επενδυτών για αυτά τα ταμεία συμπεριλαμβάνεται εδώ, όπως και στην έκθεση Σοφή. Τώρα, όσον αφορά τον δανεισμό που μπορεί να έχει ο διαχειριστής, είπαμε ότι ναι, μπορεί, αλλά δεν θα πρέπει να ξεπερνά τα ποσά των κεφαλαίων τα οποία θεωρούνται ως ε, υποχρεώσεις αλλά δεν έχουν γίνει πραγματικές πιστώσεις για να μειωθούν οι κίνδυνοι. Επίσης μίλησα για το θέμα του θεματοφύλακα. Αυτά θα πω. Νομίζω ότι δουλέψαμε πάρα πολύ επικοδομητικά και φαντάζομαι ότι θα είναι ένα θέμα το οποίο θα αποσπάσει μία εξαιρετικά μεγάλη πλειοψηφία. Προηγουμένως στο European Business Summit εξηγούσα ότι από την κατανάλωση η κινητήρια δύναμη της οικονομίας μας θα πρέπει να γίνει η επένδυση. Και πιστεύω ότι οι δύο κανονισμοί που θα εγκρίνουμε είναι κανονισμοί που μπορούν να συνεισφέρουν ταπεινά μεν, αλλά εν πάση περιπτώσει κατά κάποιο τρόπο στην ε, επανάκτηση αυτού του ισορροπίας θέλω για την οικονομία μας. Σας ευχαριστώ. Um, to... Μάλιστα, περάμε στους Κύριε Χούμπνερ, μπορούμε να ζητήσουμε πρώτα από τον κύριο Ελχαντράουι. Ευχαριστώ, Πρόεδρε, και σα ευχαριστώ πάρα πολύ που είστε έτσι ευέλικτο, γιατί θα πρέπει να φύγω σε λίγο για μια άλλη συνεδρίαση. Θα ήθελα να ξεκινήσω ευχαριστώντα ασφαλώ τον εισηγητή για το έργο και για τη συνεργασία μα. Όντω, ήταν πραγματικά εξαιρετική συνεδρίαση και στο Στρασβόργο με τους κοιόδες εισηγητές για τους συμβιβασμούς και νομίζω ότι ε, είμαστε πολύ κοντά σε μια γενική συμφωνία, σε μια συμφωνία και νομίζω ότι η έκθεση μεταφράζει πολύ σωστά αυτά που μπορούμε να πετύχουμε με τα, έργα αυτά, με τα εργαλεία αυτά για να δώσουμε μια όθηση στον τομέα αυτό γιατί αυτός είναι ο σκοπός μας να επενδύονται πιο πολύ στον, στην κοινοτομική βιομηχανία από ότι σήμερα κάποια στοιχεία, τα closed ends funds. Νομίζω ότι θα πρέπει να μεταβούμε όντως προς ένα ε, διαφανές μοντέλο και υποστηρίζει η ομάδα μου το γεγονός ότι θα πρέπει να είναι ό,τι πιο ελαφρύ γίνεται. Δεν είμαστε υπέρ του θεματοφύλακα. Καταλαβαίνω ότι ο εισηγητής θα το εξετάσει πιο προσεκτικά το θέμα αυτό. Δεν θα πρέπει να βαρύνουμε, αν θέλετε, υπερβολικά την κατάσταση και να είναι τελικά το σύστημα ε, μη ελκυστικό. Να αναφέρω επίσης ότι θα πρέπει να ε, κάνουμε μια σωστή διάκριση και σε ό,τι αφορά τις ρυθμίσεις για τα hedge funds. Νομίζω ότι αυτό συμβαίνει πολύ, με πολύ καλό τρόπο σε ό,τι αφορά τα κατόφλια. Εγώ είχα προτείνει τις 50.000 ε, ευρώ ως ε, κατόφλι, αλλά όντως θα πρέπει να υπάρχει καλή προστασία των επενδυτών, καλή ενημέρωση των επενδυτών, προκειμένου να μπορούν ενσυνείδητα να πάρουν τις αποφάσεις τους. Τελευταίο σημείο που θα ήθελα να αναφέρω και το ότι θα πρέπει το κείμενο αυτό να το συνδέσουμε και με άλλους ε, φακέλους. με το κείμενο του Ρίζοντα 2020 και με μία σειρά άλλων ε, εργαλείων επιχειρηματικότητα. Αυτά λοιπόν. Και σίγουρα νομίζω ότι η έκθεση αυτή θα υποστηριχθεί ευρέως. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ κυρία Ούμπνερ. Ευχαριστώ πολύ Πρόεδρε. Και εγώ είμαι τη ίδια άψη με του ε, συναδέλφου ότι έχουμε μια εξαιρετική συνεργασία μεταξύ σκιωδών και μεταξύ σκιωδών και εισηγήτρια. Ε, και εγώ είμαι τη ίδια άποψη ότι για τα περισσότερα ζητήματα έχουμε ήδη καταλήξει στου αναμενόμενου ε, συμβιβασμού για τι τελευταίε μικρές τροπολογίε. Πιστεύω ότι έχουμε καταλήξει σε συμφωνία σε πολλά σημαντικά ζητήματα για τους περισσότερους από εμά η επιλέξη, ο ορισμός των επιλέξιμων επενδύσεων αλλά και το ελάχιστο ποσοστό επενδύσεων καθώς και οι κανόνες που διέπουν τις διενέξεις μεταξύ εθνικών υποπτικών αρχών και πολλά άλλα θέματα και αυτό που ήταν κυρίως ε, σημαντικό για μένα καταφέραμε να συμφωνήσουμε ότι για όλα αυτά τα ταμεία που ε, αναπτύσσονται πέραν του κατοφλίου των 500 εκατομμύριων ευρώ θα συνεχίσουν να μπορούν να χρησιμοποιούν το διαβατήριο του επιχειρηματικού κεφαλαίου και πιστεύω ότι αυτή, αυτός θα είναι ένας καλός Δεν πρέπει να τιμωρούμε όσους αναπτύσσονται γρήγορα. Επίσης ήθελα να πω για αυτό το ζήτημα των 50.000 ευρώ σε σχέση με τα 100.000 ευρώ όσον αφορά το κατόφλιο εγώ είμαι διατεθειμένη να ακούσω επιχειρήματα και από τις δύο πλευρές. Καλό θα ήταν να μαζέψουμε περισσότερους επενδυτές, διότι καθαρά η Ευρώπη χρειάζεται περισσότερους επενδυτές. Από την άλλη φυσικά υπάρχουν και όλοι αυτοί οι κίνδυνοι ε, για τις ιδιωτικέ αποταμιεύσεις μια ζωή ορισμένων ανθρώπων. Αυτό θέτει λοιπόν κάποια ζητήματα και ίσως θα χρειαστεί να το ξανασκεφτούμε αυτό το ζήτημα το 50 σε σχέση με τα 100.000 ε, ευρώ για το ζήτημα του θεματοφύλακα ε, εγώ πιστεύω ότι θα πρόκειται για περιττό φόρτο για τα ταμεία που εντάσσονται στο πλαίσιο αυτού του κανονισμού. Αυτός ο κανονισμός επιχειρηματικού κεφαλαίου ε, προοριζόταν ως light καθεστώς και καλό θα ήταν να το διατηρήσουμε έτσι. Από όσο κατάλαβα, μετά από συζήτηση με συναδέλφους οι οποίες υπέβαλαν οι οποίοι υπέβαλαν τις ε, τροπολογίες υπέρ ενό θεματοφύλακα. Κατανοώ ότι ο μεγαλύτερος φόβος τους σχετίζεται με το ενδεχόμενο οι διαχειριστές ε, στο πλαίσιο της οδηγίας AFM να περάσουν στο καθεστώς ε, των κοινωνικών επενδύσεων που είναι ελαφρύτερο αλλά ειδικότερα στο άρθρο 2 αυτού του κανονισμού αποκλείονται επαρκώς ε, οι διαχειριστές αυτοί που εμπίπτουν στο καθεστώς FM ε καθώς περιορίζεται ε, το ποσό των στοιχείων του ενεργητικού κάτω από τα 500 εκατομμύρια που είναι επίσης κάτω από το κατόφλιο της οδηγίας AFM. Συνεπώς δεν βρίσκω να υπάρχουν επιχειρήματα υπέρ του θεματοφύλακα και επίζω. Ε, συμβιβασμό που προτείνει ο Φιλίπ να είναι ικανοποιητικό για όλους μας. Ε, ελπίζω λοιπόν ότι τώρα μπορούμε να επιταχύνουμε με αυτόν τον κανονισμό και αυτό θα ευχαριστήσει και τον τομέα το να μειώσουμε αυτό το διάστημα βεβαιότητας ε, καθώς μεταβαίνουμε προς αυτό το κανονισμό. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ. Ο κύριος Ντεμπάκερ, παρακαλώ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε, και από δική μου πλευρά θα ήθελα καταρχά να σα ευχαριστήσω για την καλή συνεργασία μεταξύ του εισηγητού δηλαδή και των υπόλοιπων σχεδόν εισηγητών. Νομίζω ότι αυτός ο φάκελος θα μπορούσε να είναι εύκολος αλλά και πολύ σημαντικός για τον κλάδο και νομίζω ότι θα μπορέσουμε ε, με συντριπτική πλειοψηφία να υποστηρίξουμε το θέμα αυτό. Εγώ είμαι υπέρ ενό ευέλικτου πλαισίου για το επιχειρηματικό κεφάλαιο. Θα πρέπει να δώσουμε μία όθηση στην πραγματική οικονομία. Κοιτώντας την ε, κρίση, βλέπουμε ότι υπάρχει πάρα πολύ ε, κεφάλαιο το οποίο βρίσκεται σε φάση λανθάνουσα, δεν χρησιμοποιείται και θα πρέπει να χρησιμοποιηθεί για τέτοιους σκοπούς. Ε, θέλουμε λοιπόν μία όσο πιο ελαφριά γίνεται ρύθμιση, όχι μόνο εδώ, αλλά και στην υπόλοιπη νομοθεσία σε ό,τι αφορά τα χρηματοπιστωτικά για το ευρωπαϊκό δίκαιο, ε, διαβατήριο, θα διευκολύνει ασφαλώς τις επενδύσεις και ελπίζουμε ότι θα αυξήσει και την εμπιστοσύνη των επενδυτών. Ελπίζω να αποτελέσει ε, και ένα νέο, μια νέα όθηση για το επιχειρηματικό κεφάλαιο για τους συμβασμούς τώρα που πετύχαμε στο Στρασβούργο την προηγούμενη εβδομάδα. Νομίζω ότι θα προσαρμόσουμε και θα βελτιώσουμε την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οι διαχειριστές θα μπορούν να χρησιμοποιούν το διαβατήριο ακόμα και πάνω από το όριο των 50.000 ευρώ, γιατί όχι άλλωστε, αν το σύστημα αυτό αποδείχθηκε ότι έχει επιτυχία και τα quasi equities ε, ορίζονται με καλύτερο τρόπο προκειμένου να επιτρέπονται στο Ταμείο και ο σύνδεσμος με τον ορίζοντα 2020 και με άλλα καινοτομικά εργαλεία θεωρώ ότι είναι σημαντικό. Κανά δύο σημεία μόνο παραμένουν ανοιχτά. Το depository scheme σε ό,τι αφορά τους στοματοφύλακες θεωρώ ότι αυτό το μέτρο δεν είναι θετικό, είναι δυσανάλογο. Ξέρετε φυσικά το επιχείρημα, το θέμα είναι η προστασία των επενδυτών, εντάξει, αλλά πρόκειται για άτομα συνήθως υψηλής οικονομικής επιφάνειας και γιατί δεν είναι λιανικού εμπορίου τα προϊόντα αυτά. Ξέρω ότι υπάρχουν και άλλα επιχειρήματα σε ό,τι αφορά για παράδειγμα την απόδοση κέρδους στη στιγμή που γίνεται το κέρδος αυτό. Υπάρχουν, ε, θεωρώ, πάρα πολλά επιχειρήματα που τελικά καταστούν το καθεστώς του θεματοφύλακα περιττό. Δεν είμαι πεπισμένος επίσης σε ό,τι αφορά το Key Investor Information Sheet, αυτό το φύλλο ενημέρωσης ε, των επενδυτών για μη επαγγελματίες ε, επενδυτές, μάλιστα θα μου φαίνεται λογικό, αλλά Νομίζω ότι στη σημερινή, στη, στην προκειμένη περίπτωση είναι κάτι το περιττό εφόσον απευθυνόμαστε σε επαγγελματίες. Δεν συμβάλλει ούτε στην ενημέρωση του επενδυτή, ούτε στην προστασία του καταναλωτή ιδιαίτερα. Θεωρώ όμως ε, συνολικά ότι τα δύο βασικά θέματα τα οποία παραμένουν ανοιχτά ε, για τα θεματοφύλακα και για το Key Information Investors Sheet είναι τα δύο νυχτά ζητήματα στα οποία θα καταλήξουμε σε μια συμφωνία πολύ σύντομα προκειμένου να μπορέσουμε να δώσουμε μια νέα όθηση, όπως είπα, στα, κεφάλαια, στα, κεφάλαια, στα επιχειρηματικά κεφάλαια. In which case then uh, the rapporteur would like to conclude. Ε, Δεν έχω πολλά να προσθέσω. Αυτό που θα κάνω είναι θα επεξεργαστώ και θα εντάξω αυτά τα δύο σημεία τα οποία παραμένουν ανοιχτά μέσα στην έκθεση. Μέσα σε μία εβδομάδα λοιπόν θα σας έχω διαβιβάσει τα καινούργια κείμενα για να μπορέσουμε να συζητήσουμε αυτά. Μάλιστα λέει ο Πρόεδρος. Προθεσμία για κατάθεση τροπολογίων τέλη Μαΐου, 31 Μαΐου και μετά θα δούμε πότε θα ψηφιστεί τον Ιούλιο ή όχι στην Ολομέλεια. Το επόμενη συνεδρίαση, η Δευτέρα 7 Μαΐου, 3 το απόγευμα. Και θα ακολουθήσει και άλλη συνεδρίαση την Τρίτη στις 8 Μαΐου στις 9 το πρωί. Ευχαριστώ πολύ. Πέρα στη συνεδρίαση.